Περιμένουμε ακόμα κάποιου ευρωβουλευτέ. Δεν θα περιμένω άλλο, Όμω ε, ήδη είναι 9 και 6. Καλημέρα σε όλου. Α ε, σας παρουσιάσω πρώτα τα αποτελέσματα από τι συνεδρίε των ε, συντονιστών. Καταρχά υιοθετήθηκε η ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου. Όσον αφορά τις ε, έκθεσεις και γνωμοδοτήσει, παρακαλώ η πίσω δεξιά να είστε λίγο πιο ήσυχοι. Εκθέσεις και γνωμοδοτήσει. Ο κύριος Βαλένσα από το ΕΛΚ έχει αναλάβει τον ε, κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών όσον αφορά την παρακολούθηση τη εφαρμογή ε, τη της Ευρωπαϊκής και των πίνακα αποτελεσμάτων. Έχουμε αναβάλει τις αποφάσεις αυτές ε, από ε, τις επίμαχες συστάσεις. Είχαμε ένα ε, αίτημα για τις αναφορές σε 5.99 και 6.17 από το ΕΛΚ και, το, και τους σοσιαλιστές αντίστοιχα. Η 604 αναβλήθηκε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση και οι επόμενες εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις δικές μου συμβαστικές προτάσεις. Η διαρευνητική επίσκεψη στην Λουσατία παρουσιάστηκε με αναθεωρημένο πρόγραμμα. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή για την επίσκεψη αυτή. Τέσσερα μέλη μπορούμε να δεχτούμε ακόμα, δύο εξοφίκιο και δύο πλήρη μέλη. Θα πρέπει όμως να ε, δηλώσετε το ενδιαφέρον σας πριν τις 27 Νοεμβρίου. Επίσης, ζητήσαμε από τον Προεδρείο να ε, μεταφράσουν τα παραρτήματα ε, της έκθεσης της Ομάδας Εργασίας ε, για την Ευμερία των Παιδιών. Αποφασίστηκε να ζητήσουμε μετάφραση στα γαλλικά και γερμανικά μόνο, εφόσον το αγγλικό κείμενο ήδη υπάρχει. Γαλλικά και γερμανικά είπα, λέει η Πρόεδρος. Στα γαλλικά και γερμανικά θα, μεταφραστεί, θα μεταφραστούν τα παραρτήματα όσον αφορά τις ε, μελέτες ε, του ε, θεματικού τμήματος και για τα εργαστήρια. 27 Νοεμβρίου, 10 η ώρα το πρωί είναι η προθεσμία την υποβολή προτάσεων. Κατόπιν έχουμε την ΦΑΤΚΑ, την αναφορά υπαριθμών 1088. Αποφασίσαμε να στήσουμε από το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ σχετική μελέτη. Περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περιμένουμε μέσα Ιανουαρίου. Στο μεταξύ, οι συντονιστές θα εξετάσουν περαιτέρω δράσεις σε πολιτικό επίπεδο στις συναντήσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Αποφασίσαμε να υποδεχτούμε για σύντομη επίσκεψη το Μαροκινό Κοινοβούλιο χωρίς ανταλλαγή απόψεων. Πρόκειται απλά για μια επίσκεψη εθιμοτυπίας και, θα θέλουμε να αναθεωρήσουμε ε, τις προθεσμίες ε, για την υποβολή ετοιμάτων ε, για κατατμήματα και χωριστές ψηφοφορίες. Η νέα προθεσμία τώρα είναι δύο μέρες πριν την ψηφοφορία το μεσημέρι. Τίποτα άλλο. Προχωράμε τώρα. Everything has happened. That was a... τι να πω, πολύ ωραία μουσική τώρα. Μόλις με ενημερώνουν ότι οι αναφέροντες δεν βρίσκονται στην αίθουσα, τους, παραμένουμε ακόμα. τους περιμένουμε ακόμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Hm. So where did the music come from? Was Η μουσική από πού προήλθε, από το τηλέφωνο κάποιου. Wow, but let's enjoy the music Ας απολαύσουμε τη μουσική στο μεταξύ. je pense que ce n'est pas de la musique, c'est l'accompagnement d'un film qui doit être projeté pour la pétition suivante. Δεν είναι μουσική, είναι η συνοδεία μια ε, ταινία, ε, είναι μάλλον η μουσική υπόκριση μια ταινία η οποία ε, είναι τμήμα τη παρουσίαση του επόμενου θέματο. So, thank you very much for being here very early. Ευχαριστώ που ήρθατε τόσο νωρίς εδώ. Είναι η αναφορά 37, σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Ε, αν συμφωνείτε μπορούμε να συζητήσουμε πρώτα αυτό το θέμα. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επομένως μπορούμε ε, να επιδείξουμε πρακτικό πνεύμα και να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα στη διάθεσή μας. Ε, αναφορά 37 για την κατασκευή ενός μεγάλου αυτοκινητοδρόμου περιφερειακού γύρω από την πόλη της Ορλεάν. Ο αναφέρον, ο κύριος Ζων Μαρή Σαλωμόν είναι εδώ μαζί ε, ίσως και με το σύμβουλό του και να σας δώσω απευθεία το λόγο. Έχετε και μία μικρή ταινία. Πολύ ωραία.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 maybe Ίσως ε, θα έπρεπε λίγο να εξηγήσω ότι οι Ισπανοί που είναι εδώ για το προηγούμενο θέμα μπορεί να ενοχληθούν λίγο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν είναι εδώ οι αναφέροντες. Προκειμένου λοιπόν ε, να μην χάσουμε άλλο χρόνο, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Να δώσω λοιπόν το λόγο στο Ζαμαρί Σαλομών και να σας πω ότι έχετε και δύο λεπτά ακόμα αν θέλετε να εξηγήσετε περισσότερα για το θέμα. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, μιλώ εξ ονόματος 220 μελών της Ένωσης Μάρτιε Είμαι πρόεδρος και σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Συνοδεύομαι από τον κύριο Σολέρ, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της Ένωσης ε, και είναι και ερετό μέλος ε, της περιοχής του Λουαρέ. Το Λοαρέ ε, στην, ε, στα νότια του Παρισιού διασχίζεται από το Λίγυρα, το πιο μεγάλο ποταμό που είναι ακόμα, ε, έχει ακόμα άγρια φύση στην Ευρώπη. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια προσπαθούν στην περιοχή της Ορλεάνης να επιβάλλουν μια παράκαμψη 15 χιλιόμετρων που περιλαμβάνει και μια γέφυρα 600 μέτρων πάνω από το Λίγυρα. Ε, πρόκειται για ένα ε, χώρο ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη βιοπικιλότητα ε, και είναι και περιοχή ε, της UNESCO. Έχει ταξινόμηση GPS και GSE Natura 2000, καθώς επίσης και προστατεύεται από άλλη γαλλική νομοθεσία. Παρά το ψήφισμά σας στις 23 Σεπτεμβρίου του 2008, που κατήγγειλε τον κίνδυνο παραβιάσεων των οδηγιών Habitat και των οδηγιών για τα πουλιά. Το έργο συνοχίζεται και πέρσι ε, δόθηκε έγκριση από μία δήλωση ε, ε, χωροταξίας του εισαγγελέα της περιοχής του Λουαρέτ. Υπάρχει η οδηγία 9243 που αναφέρεται στο άρθρο 6 ότι θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα για τη διατήρηση ειδών και την, το ενδιαίτημά τους και επομένως θα έπρεπε να βρεθούν κάποιες άλλες λύσεις οι οποίες αγνοήθηκαν οι επιθέσεις στο περιβάλλον θα είναι πάρα πολύ σοβαρές, διότι προβλέπεται ε, <clears throat> ότι θα ε, χαθεί ένα τμήμα πρασίνου για αστικοποίηση της περιοχής της Ορλεάνης. Υπάρχει εξαιρετική βιοπικιλότητα, πάνω από 150 είδη άγριων πουλιών, πάνω από 30 είδη λιβελούλες, 9 ε, είδη νυχτερίδας ε, και φυσικά και πανίδα και χλωρίδα, συγγνώμη. Ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές οι συνέπειες ε, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, η ε, εκτίμηση επιπτώσεων δεν λαμβάνει υπόψη της τα 74 είδη τα οποία είναι προστατευόμενα από το παράρτημα 1 της οδηγίας για τα πουλιά. Μπορεί να υπάρξει καταστροφή ή διαταραχή των συγκεκριμένων ειδών στην περιοχή ή να υποβαθμιστεί ο χώρος αναπαραγωγής τους και διαβίωσής τους και δεν λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο ε, κάποια ε, ισχνά ε, θετικά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Από το 1996 το έργο προβλέπεται λόγω της πρόβλεψης ότι θα αυξηθεί η οδική κίνηση. Αντίθετα όμως διαπιστώνεται ότι έχει υπάρξει μείωση της κίνησης στην γέφυρα του Ζαργό και είμαστε στο 80% της προβλεπόμενης κίνησης. Ε, το ε, σχέδιο δεν φαίνεται ότι θα μειώσει τα προβλήματα της κίνησης, αλλά αυτοί οι οποίοι παρακάμπτονται και πηγαίνουν σε ε, κοντινές περιοχές ε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα, να υπάρχουν περισσότερες συνοχλήσεις, περισσότερα ατυχήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η παράκαμψη δεν θα βοηθήσει ε, καθόλου βάσει των προβλεπόμενων μεγεθών. Δεν εξετάστηκε ποτέ μια εναλλακτική λύση και υπάρχει και απηγή ε, τη δημιουργία, για παράδειγμα, ε, μιας ε, ε, Ενό σταυροδρόμιου κάπου εκεί κοντά, να υπάρξει συντανισμό των ε, ωραρίων ε, των εργοστασίων που βρίσκονται στην περιοχή. Ζητάμε λοιπόν να γίνει αναθεώρηση αυτού του σχεδίου, το οποίο θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την περιοχή και θα ήθελα να σας ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι ευρωπαϊκές οδηγίες και να εφαρμοστεί πολύ σύντομα ένα σχέδιο το οποίο θα σταματήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Je vous remercie. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στον κύριο Σπάικτ. Merci. Η Κομισιόν έλαβε γνώση αυτής της ενημερωμένης αναφοράς που αναφέρεται στον αντίκτυπο ε, του ενός ε, σχεδίου σε ένα χώρο Natura 2000 οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τηρηθεί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω τις διάφορες διαδικασίες και τα διάφορα στάδια. Υπ' αυτή την ε, έννοια η Κομισιόν θεωρεί ότι καταρχήν οι ενώσεις οι αναφέροντες θα πρέπει να προσφύγουν καταρχήν στην εθνική δικαιοσύνη. Κοινού δικαίου δηλαδή για την εφαρμογή τη ε, νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, το έχουν ήδη κάνει. Παράλληλα, μια και το σχέδιο αυτό ε, θα επηρεάσει διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, η Κομισιόν μπορεί να εξετάσει τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία ε, κοινοποιούνται από το κράτος μέλο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της ε, οδηγίας για τα οικοσυστήματα. Και θα μπορούσαμε ενδεχομένω να ζητήσουμε και διευκρινήσει από τις γαλλικέ αρχές. Επί τη ουσία, οι αναφέροντες ε, αναφέρουν πως το σχέδιο δεν ε, σέβεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το από τα σχέδια ε, γενικού ενδιαφέροντος, καθολικού ενδιαφέροντος. Όμως, το σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας και την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Είναι στόχοι αξιόλογοι. Τώρα, τίθεται ενδεχομένω θέμα αναλογικότητας. Και πάλι, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν τα εθνικά δικαστήρια. Κατά συνέπεια, η Κομισιόν δεν έχει εντοπίσει συγκεκριμένους λόγους που θα δικαιολογούσαν την παρέμβασή τη, οπότε καλεί τους αναφέροντε να συνεχίσουν τη δράση τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές. Και να θυμίσω σε όλους ότι πρόκειται για μία αναφορά που είναι ανοιχτή εδώ και 12 χρόνια. Είναι λοιπόν πολύ περίεργο που ο χρόνος ε, τρέχει και δεν φαίνεται κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Μαρκρέτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμετείχα σε διευρυντική επίσκεψη στην περιοχή αυτή πριν πολύ καιρό. Τουλάχιστον πριν πέντε χρόνια. Ήταν όμως ήδη τότε σαφές ότι τα σχέδια για αυτόν τον αυτοκινητόδρομο σε αυτήν την ε, καταπληκτική περιοχή ε, δεν ε, ήταν παρκώς αιτιολογημένα. Δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση τώρα. Υπήρχε όμως δρόμος με διόδια και επειδή ε, είχε διόδια, δεν ε, είχε συμπεριληφθεί στα σχέδια των μεταφορών στην περιοχή αυτή. Και γι' αυτό θεωρήθηκε ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέος δρόμος. Ε, δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, δεν είχα το χρόνο να το εξετάσω αυτό αναλυτικά, αλλά... Φαινόταν ότι δεν υπήρχε επαρκής λόγος να δημιουργηθεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος από τις αρχές και τη στιγμή που δεν γίνεται τίποτα, υπάρχει τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θέλω να κανέναν, κανέναν, ε, να μην αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Και έτσι ε, έχουμε αυτές τις ε, συνεχείς post-mortem αντιδράσεις εδώ στην Επιτροπή μας τις αυτοψίες, να το πούμε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, διότι είναι μια σαφής απειλή σε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Ε, να θυμίσω σε όλους, λέει η Πρόεδρος, ότι το 2007 πραγματοποιήθηκε η διερευνητική επίσκεψη, πριν 10 χρόνια. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, Ελεονόρα. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφο Σάουκεν. Θεωρώ ότι η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, διότι παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια ε, και είναι ακόμα ανοιχτή, είναι σαφές ότι από τη μια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ακλόνητη και οι τοπικές αρχές όμως, οι οποίες ε, καθυστερούν και εξακολουθούν να αγνοούν πάρα πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα τα οποία παρουσίασαν οι αναφέροντες, διότι νομίζω ότι η ουσία εδώ είναι αυτή. Κάποιες πολιτικές, ιδίω σε θέματα βιωσιμότητας, εξακολουθούν να κλείνουν το μάτι σε ένα μοντέλο που βασίζεται στο ε, τσιμέντο, στην βιωσιμότητα μέσω των οδικών μεταφορών, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν πιο ευέλικτα μοντέλα το 2017 και αυτές είναι οι σωστές επενδύσεις, όχι μια επένδυση η οποία θα διαταράξει μια τόσο όμορφη περιοχή. Εάν θέλουμε λοιπόν να στείλουμε άλλη μια επιστολή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπής μα μάλλον, συγγνώμη, θα μπορούσαμε ίσω να κάνουμε κάτι ακόμα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Thank you. Peter, Ο Πέτερ Γιάρ. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση και μια συγκεκριμένη. Η γενική μου παρατήρηση είναι ότι γενικά συχνά έχουμε επικρίνει σε τέτοια μεγάλα έργα στα αρχικά στάδια του προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προϋποθέτει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ε, τηρήσουν ε, τους κανόνες και έτσι θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εγώ νομίζω ότι ήδη στις αρχικές φάσεις θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένας επικοδομητικός διάλογος, να το ονομάσω έτσι και αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ε, έχουν γίνει όλα σωστά ή όχι. Εμένα μου λείπει αυτό, ένας διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική φάση, διότι σε πολλές περιπτώσεις ε, τότε μπορεί να γίνουν κάποιες διορθώσεις και μάλιστα με αμοιβαία συνένεση. Θα ήθελα να συστήσω στον αναφέροντα να εξαντλήσει τις ε, δικαστικές δυνατότητες ε, στην ε, Γαλλία. Σε αυτό συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να εξαντληθούν δηλαδή οι δυνατότητες προσφυγής εντός της χώρας. Δεν ξέρω, έχουν εξαντληθεί, έχουν ξεκινήσει, τι ακριβώς γίνεται, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω την αναφορά όχι επειδή είμαι ικανοποιημένος με την πορεία των πραγμάτων, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω, πρέπει να κινηθούν δικαστικά οι αναφέροντες. Η ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Είναι τόσο παλιά αυτή η υπόθεση που ε, ε, δεν ε, ήμουν να καν ευρωβουλευτή στην Επιτροπή αυτή όταν ξεκίνησε. Αλλά βλέπω να υπάρχει μια πολύ θλιβερή τάση σε διάφορες υποθέσεις που θα συζητήσουμε τώρα το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιδρά με στεναρό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με τους συναδέρφους μου ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Όκεν, ε, ναι, συγγνώμη, επειδή ε, σκεφτόμουν πολύ τη δανέζικη υπόθεση, ε, δεν είχα συνειδητοποιήσει το εξή και μόλι τώρα με ενημέρωσαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτή είναι η καινούρια στρατηγική τη Επιτροπή, είναι στην στο περιβάλλον ασχολείται με μικρά πράγματα. Δεν είναι οικονομικό θέμα και γι' αυτό δεν ασχολείται. Ξέρω ότι αυτή δεν είναι η θέση τη Γενική Διευθύνση Περιβάλλοντο. Ε, είναι όμω ε, τμήμα τη ε, στρατηγική για την βελτίωση τη νομοθεσία. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφεύγει να ε, προχωρήσει σβάθος σε υποθέσεις ε, που παραβιάζουν το περιβαλλοντική νομοθεσία. Και αυτό φαίνεται από ό,τι γνωρίζω στην τελευταία απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε σε εθνικό επίπεδο, δεν χρειάζεται να ανακατευτούμε εμείς. Θα θυμάστε ο Τίμερμανς ε, που προσπάθησε να καταστρέψει την οδηγία ε, για την ε, Natura. Δεν τα κατάφερε και ευτυχώς. Ε, αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την περιβαλλοντική νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να γίνει, παρότι οι παρόντες μάλλον δεν είναι υπεύθυνοι. Ε, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, αραιώνει, να μην αποδυναμώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλου ομιλητέ εδώ πέρα. Να ξαναδώσουμε το λόγο στου αναφέροντε για να συνοψίσουν και για να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν, έχει, αν έχετε μετακινηθεί στις Παρακαλώ, δύο λεπτά έχετε. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω σε από τα σχόλια που άκουσα. Το σχέδιο αυτό ε, χρονολογείται ε, από εδώ και 20 χρόνια στην πραγματικότητα. Γιατί το Νομαρχιακό Συμβούλιο προσπάθησε και άλλες εναλλακτικές ε, λύσεις οι οποίες όμως δεν έδωσαν αποτέλεσμα. Οπότε ζητούμε ξανά από το Κοινοβουλίο να τοποθετηθεί, διότι το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε ξανά εδώ και ένα χρόνο περίπου και μπαίνει στη φάση έναρξης ε, των ε, εργασιών. Έχει ήδη γίνει εκρίζωση δέντρων, ένα κομμάτι του δάσους καταστράφηκε ήδη και προφανώς θα ε, ξεκινήσει τώρα, θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, αλλά ήδη βρισκόμαστε στη φάση έναρξης. Η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να προσφύγουμε ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Το έχουμε κάνει εδώ και ένα χρόνο. Αλλά ακόμα δεν μα έχουν δώσει ημερομηνία για μια πρώτη ακρόαση σε πρώτο βαθμό. Οπότε αν υπολογίσουμε και τις ενδεχόμενες προσφυγές φοβόμαστε ότι το έργο θα έχει τελειώσει πριν ακόμα η γαλλική δικαιοσύνη τοποθετηθεί επί της νομιμότητάς του. Η δήλωση δημοσίου συμφέροντος ε, ε, ε, είναι αντιφατική, δε, κρύβει μια σύγκρουση συμφερόντων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα γενικό ενδιαφέρον για το έργο από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά μια βλάβη στο περιβάλλον που θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογα μεγάλη για τα κέρδη για, για τα ωφέλη μάλλον που θα προκύψουν από το έργο αυτό. Και θα θέλαμε και εσείς να ζητήσετε από την γαλλική κυβέρνηση να επιβεβαιώσει αυτά που λέμε, να αναλάβει δράση, να μην αφήσει την τοπική αυτοδιοίκηση Γαλλίας, ε, την τοπική αυτοδιοίκηση στο Λίγυρα να προχωρήσει αυτό το έργο. Πρόεδρος, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, εκρεμεί εδώ και 20 χρόνια και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Ευχαριστούμε πολύ για τους αναφέροντες που απευθύνθηκαν σε εμά. Είναι ένα θέμα το οποίο πηγαίνω έρχεται. Είναι προφανώς ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αν δούμε την οδηγία Natura 2000, για παράδειγμα, το άρθρο 6 παράγραφος 4 για τα οικοσυστήματα. Ε, το καταλαβαίνουμε, είναι ένα θέμα συνολικό ευρωπαϊκό θέμα, όχι μόνο γαλλικό. Δεδομένου το θέμα όμως ε, στα γαλλικά δικαστήρια αυτή τη στιγμή, η Κομισιόν αποφάσισε ότι θα πρέπει το γαλλικό δικαστήριο να αποφανθεί πρώτα. Εγώ από την άλλη μεριά προτείνω να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε να υπογραμμίσουμε ε, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το γεγονός ότι είναι θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ε, το γεγονός ότι ενδεχομένως υπάρχει θέμα σύγκρουση συμφερόντων, αλλά θα πρέπει να καλέσουμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, και ιδιαίτερα στις γαλλικές αρχές. Οπότε θα πρότεινα να στείλουμε μια επιστολή στις γαλλικές αρχές, υπενθυμίζοντάς τους ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού κατά την εφαρμογή των οδηγιών που υφίστανται και να τους υπογραμμίσουμε τη σύγκρουση ε, μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και της ε, περιβαλλοντικής ζημίας. και, αλλά και πιστεύω ότι ε, μέχρι να μα απαντήσουν οι γαλλικές αρχές δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αφορά. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρουμε ρητά ότι χρειαζόμαστε επιγόντω μια γραπτή απάντηση. Μια και το θέμα εκκρεμεί σε γαλλικό δικαστήριο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάργαρετ. Συγγνώμη που δεν είμαι επαρκώ προετοιμασμένη, ζητώ συγγνώμη, αλλά... δεν υπάρχει μια μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις γαλλικές αρχές. Και δεν μπορούμε να δούμε το κατά πόσον οι συστάσεις που είχαμε εκδώσει μετά την διαρευνητική μας αποστολή υλοποιήθηκαν. Γιατί η Κομισιόν είναι τόσο αόριστη σε αυτά που λέει. Θα τις χάσουμε όλες αυτές τις υποθέσεις. όπως και την επόμενη. Κατόπιν εορτής θα έρχονται και θα λένε εντάξει πέθανε ο ασθενής αλλά ε, δεν έγιναν σωστά τα πράγματα. Τι να το κάνουμε. Πρόεδρος, συμφωνώ. Πίτερ, έχεις και εσύ το λόγο. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι. που με θυμώνει κάπως. Θα προτιμούσα να είναι εδώ οι παρόντες οι Γάλλοι συνάδελφοι. Κάτι που με ενοχλεί λίγο όσον αφορά τη δικαστική οδό. Ε, συνήθως ε, σε αυτές τις ε, περιπτώσεις ο δικαστής λέει ότι δεν έχει νόημα να παρέμβω αν έχει ήδη το το έργο. Εάν λοιπόν ακολουθήσει κανείς ε, την ε, δικαστική οδό θα πρέπει καταρχάς ε, να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου. Μήπως να ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Θα πρέπει πριν ξεκινήσει το έργο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Ε, δεν μου ακούγονται πολύ καλά τα πράγματα. Το λέω αυτό με μη νομικούς όρους. Δεν είμαστε δικαστήριο. Μπορούμε όμως να πούμε ότι αν είναι σωστά αυτά που μας έχουν πει οι αναφέροντες, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Ε, αν ε, υπάρχει η δυνατότητα παρέμβαση, έχει καλώ. Αλλά αλλιώ ε, τι θα γίνει, θα πούνε ότι τώρα ολοκληρώθηκε το έργο και άλλωστε οι αναφέροντες δεν θέλουν χρηματική αποζημίωση, θέλουν το έργο αυτό να συμπορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τους συναδέρφους, να το συμπεριλάβουμε αυτό στην επιστολή προς, ε, τους, ε, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, πρόεδρος. Πίτερ, δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ρωτάμε τους ε, συναδέρφους. Είναι μια υπόθεση που εκκρεμεί στο δικαστήριο, για όνομα του Θεού. Να στραφούμε στις γαλλικές αρχές, να ζητήσουμε μελέτη επιπτώσεων να ζητήσουμε κατά πόσο συμμορφώνεται με τις δύο ισχύουσες οδηγίες το έργο αυτό και να ζητήσουμε επιγόντως να μας υποβάλουν γραπτή απάντηση εδώ στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνείτε? Εξαιρετικά. Ευχαριστώ τους αναφέροντες. Γνωρίζετε τώρα ότι παρακολουθούμε το θέμα, θα απευθυνθούμε στις ε, γαλλικές αρχές ε, και θα τους ε, επισημάνουμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, θα πρέπει όμως να ενεργήσουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα στην προηγούμενη αναφορά, την αναφορά 2582 για το τρένο υψηλή ταχύτητα μεταξύ Μαδρίτης και Μούρθια. Νομίζω ότι είναι παρόντες τώρα πια οι ε, αναφέροντες. Σας καλωσορίζω θερμά. Έχουμε επίσης την αναφορά 19 σχετικά με το υπόγειο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλή ταχύτητα στην πόλη Μούρθια. Ε, και αυτός ο αναφέρον είναι παρόν. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Κοντρέρα Ριβέρα και στην αναφέρουσα που προτιμάει να είναι ανώνυμη. Πέντε λεπτά ο καθένας, παρακαλώ. Buenos Καλή σας μέρα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που στρέφετε το βλέμμα σας στην περιοχή μας και στη Μορφιά σας χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε δώσει μάχη έτσι ώστε το τρένο υψηλής ταχύτητας προς τη Μούρθια να είναι υπόγειο. Το 1991 πετύχαμε και το 1995 ε, Επίση, το 2006 μια, ε, καταλήξαμε μια συμφωνία που υποχρέωνε την υπογειοποίησή του. Έτσι έγινε και η εκτίμηση περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων το 2009. Η κυβέρνηση όμως περιόρισε ε, το έργο ε, σε, ε, και ζήτησε να γίνει υπέργειο. Μετά από χρόνια αντιδράσεων έγινε δεκτό το αίτημά μας έτσι ώστε η υπογειοποίηση να γίνει αλλά περιορίζεται στα 1100 μέτρα απομένουν άλλα 5,5 περίπου χιλιόμετρα για να καλυφθούν να γίνουν, σεβαστή η να γίνουν σεβαστοί περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε επανειλημμένο στην Ισπανία για την συστηματική παράβαση τη ε, κοινοτική νομοθεσία ε, περιβαλλοντικού κινδύνου μέσω, για παράδειγμα, κατακαιρματισμού ε, των έργων που έχουν περιβαλλοντικό κίνδυνο. Κάτι παρόμοιο έγινε και στη Μούρθια. Μάλιστα, είναι αδύνατον να ζητήσουμε την παράλυση του έργου για περιβαλλοντικούς λόγους. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τον εισαγγελέα περιβάλλοντος να κάνει μια προσφυγή και το έκανε. Εξαιτία όμως της ε, Ισπανικής νομοθεσία δεν του αναγνωρίστηκε νομιμοποίηση αν το κάνει. Η αρμοδιότητα δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Ε, το έργο αυτό παραβιάζει ε, την ε, κοινωνική νομοθεσία και ιδιαίτερα τη σύμβαση του Άρχους. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στα έγγραφα τα οποία σας υποβάλαμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι η δική μου κατάσταση, καθώς επίσης και άλλων χιλιάδων γειτόνων μου. Ε, ζω σε μια ζώνη εκτός της υπογειοποίησης των 1100 μέτρων. Ζω σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα σχέδιο. Το μόνο που υπάρχει είναι μια ε, απόφαση, κυβερνητική απόφαση, που επιτρέψει το τρένο να περάσει υπέργεια. Ε, ε, αυτή είναι μία από τις υπόγειες διαβάσεις ε, για τους πεζούς που παλιά χρησιμοποιούσαν μόνο οι ροϊνομανείς. Ε, είναι, από εκεί θα πρέπει να περνάμε για να διασχίζουμε τις ε, γραμμές. Ε, είμαστε καταδικασμένοι να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους υπόγειες διαβάσεις πεζών. Εμείς το χρησιμοποιούμε χιλιάδες φορές το χρόνο. Εμείς, τα παιδιά μας για να πάνε στα σχολεία, στο κέντρο υγείας, στην εκκλησία και από εκεί θα πρέπει να περνάμε επιστρέφοντας μόνες μας στο σπίτι μας ε, το βράδυ και οι δικοί μας να μας περιμένουν ανήσυχοι μέχρι να ακούσουν το κλειδί στην πόρτα. Είναι... Ε, ε, έχουμε δει πόσες φορές έχουμε, έχει γίνει παραβίαση των, των, ε, της, της νομοθεσίας, της νομοθεσίας γι' αυτό. Ε, είμαστε χιλιάδες που δεν θέλουμε την πόλη μας διαρεμένη στα δύο. Είμαστε χιλιάδες αυτοί που θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας και μερικές φορές και για τα εγγόνια μας. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι το τρένο υψηλής ταχύτητα θα έπρεπε να φτάσει υπογειοποιημένο στο σύνολό του. Αλλά μας είπαν ψέματα και θα μας το φέρουν έτσι, όπως το βλέπετε εδώ. Γι' αυτό το λόγο σας ζητούμε να μην κλείσετε την αναφορά αυτή. Κάντε ό,τι μπορείτε. Ε, ξεκινήστε μια διαδικασία ε, κάντε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε οι εισαγγελείς να μπορέσουν να προστατεύσουν τους ε, πολίτες, να υφίσταται στην πραγματικότητα η διάκριση μεταξύ των εξουσιών. Ε, μη μας αφήσετε μόνους μας. Ε, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για ένα υπογειοποιημένο τρένο θα πρέπει να ελοπιθούν. Μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο, συγγνώμη, το δεύτερο εκ των αναφερομένων. Έχετε το λόγο για άλλα πέντε λεπτά. Αξιότιμοι κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ε, εδώ και 30 χρόνια συνεχίζεται η διαδικασία. Έμειναν πίσω 10 σύντροφοι με τους οποίους ε, ξεκίνησα τη μάχη, όπως ο πατέρας Τορνέλο, ο οποίος ήταν ε, σύντροφός μου στη μάχη και ε, χάθηκε από τον καρκίνο χωρίς να ζήσει το όνειρό του, να υπάρχει αυτό το υπόγειο τρένο. 30 χρόνια υποσχέσεων οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Όταν υπεγράφει η σύμβαση για το υπόγειο τρένο πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε πετύχει τα πάντα. Τα πράγματα δεν πήγαιναν άσχημα. Το 2009 εγκρίθηκε και η εκτίμηση περιβαλλοντικών υποπτώσεων και έγινε μεταρρύθμιση του σχεδίου χωροταξία. Αλλά μετά το 2012 εγκρίθηκε ένα πρώτο σχέδιο το οποίο έγινε δεκτό το 2012 για να γίνει υπέργειο το τρένο. Έκτοτε βρισκόμαστε στο δρόμο. Ε, κάθε Τρίτη ε, γίνονται διαδηλώσει ε, και φτάσαμε και στη μεγαλύτερη διαδήλωση που έζησε η περιοχή τη Μούρσια κάποια Σήμερα Έχουμε 73 συνεχείς ημέρες ε, όπου 20 με 23 μέρες βρίσκονται ε, χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο στη Μούρθια. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Μόνο όταν η Ευρώπη θα μπορέσει να ρίξει μια ματιά στο τι συνέβη, ε, άρχισε να δράει η Ισπανική κυβέρνηση. Στην αρχή για να έχουμε 30 μέτρα, μετά άλλα 580 μέτρα κάτω από τη γη και έχουμε 1100 ε, μέτρα τα οποία είναι λιγότερα από τα 1800 υπόγεια που μας στα 7-800 συγγνώμη που μας είχαν υποσχεθεί. Καταγγείλαμε αυτή την παρανομία σε κάθε περίπτωση και στις ε, υπηρεσίες περιβάλλοντος, ε, οι οποίες ε, ε, διαπίστωσαν ότι ο Ισπανικός νόμος ε, ε, δεν καλύπτει την Ευρωπαϊκή Οδηγία και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοποίηση. Πήγαμε στον Ισαγγελέα υπεύθυνο για θέματα περιβάλλοντος. Το καταγγείλαμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κάναμε και στο παρελθόν στο Δήμο της Μούρθια, ο οποίος έκανε μια μελέτη και διαπίστωσε ότι υπάρχει πιθανότητα παρανομίας, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μόνο όταν φτάσαμε εδώ, καταγγείλοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, ότι έχει αλλάξει ε, και ότι υπάρχουν θέματα περιβαλλοντικά τα οποία δεν έχουν επιληθεί, μόνο τότε η Ισπανική κυβέρνηση άρχισε να κάνει κάποια βήματα. Γι' αυτό ακριβώ σα ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Σα παρακαλώ, μελετήστε όλα όσα πρέπει να μελετηθούν, ε, δείτε τι γίνεται και να κινήσετε όλα τα νήματα προκειμένου να σταματήσει αυτή η τρέλα για να μην συμβεί κάτι τέτοιο οπουδήποτε αλλού. Το τρένο υψηλή ε, ε, είναι όλο και πιο κοντά στην υπέργεια κατασκευή του. Και η πόλη θα διαιρεθεί στα δύο και οι γειτονιές μας ε, θα είναι εκτός της πόλης. Στην περιοχή στην οποία ζω εγώ σήμερα δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Υπάρχουν μόνο ε, υποσχέσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή Εάν ε, το τρένο γίνει υπέργειο, δεν θα έχει καμία σχέση με το σχέδιο του 2006. Θα χωριστούν γειτονιέ και οι οικογένειε οι οποίε ζούσαν σε απόσταση 5 λεπτών τώρα θα πρέπει να πάρουν αυτοκίνητο για να συναντηθούν. Και ε, νομίζω ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν υπάρχει ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν θυσίε, αυτό το δεχόμαστε, αλλά ε, αν είναι για να έχουμε ένα τρένο υπόγειο, τότε αξίζει τον κόπο. Αλλά δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν ένα υπέργειο τρένο, το οποίο είναι αντίθετο από αυτά που συμφωνήθηκαν. Σήμερα στη Μούρθια δεκάδες χιλιάδες γειτόνων κοιτούν προς την Ευρώπη. Δεν μπορούν να έρθουν. Είναι άνθρωποι ταπεινοί, αλλά με αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια που του ζητούσε ο πατέρας Τορνέλ. Θέλουν ε, Είναι οικογένειε που δεν θέλουν να χωριστούν από την πόλη. Θέλουν να συμμετέχουν στο όνειρο που του υποσχέθηκαν κάποια στιγμή. Είναι δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι που δεν θέλουν να δουν ε, ότι τα παιδιά του, ε, αγόρια και κορίτσια, περνούν από γειτονιέ και μπορεί να ξεχαστούν αυτά τα πράγματα τα οποία του υποσχέθηκαν κάποια στιγμή. Ελπίζουμε λοιπόν να μην συνεχιστεί αυτό το τρένο υπέργειο, διότι θα χαθεί αυτό το όνειρο. Ε, Μόνο την νομοθεσία, δεν τηρούνται αυτά τα οποία ε, μας υποσχέθηκαν. Έχουμε κουραστεί, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή η Επιτροπή θα διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά μας για να υποχρεώσει το Ισπανικό κράτος για ε, να τηρήσει μια φορά ε, την υπόσχεση που μας έχει δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, yes, many thanks. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά αυτή είναι πολύπλοκη. Ε, έχει να κάνει με την ε, οδηγία εκτίμησης περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων. Έχει να κάνει με τα τούνελ κάτω από την Μούρθια. και το 2014 ε, φάνηκε να τροποποιείται το έργο αυτό. Και στείλαμε επιστολή τότε στις ε, Ισπανικές Αρχές ε, και τους είπαμε ότι όταν αλλάζει κανείς σε σημαντικό βαθμό ένα έργο θα πρέπει να, ξανα... να έχουμε μια νέα μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και Τότε, το 2015, οι Ισπανικές αρχές ε, επιβεβαίωσαν ότι όχι, θα συνεχίσει να ισχύει η αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν υπήρχε ε, παραβίαση του νόμου. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο στοιχείο που είχαμε στα χέρια μας, ε, ωστόσο τώρα ακούμε και πάλι από τους αναφέροντες αυτά που λένε. Θα εξετάσουμε τους ισχυρισμούς αυτούς και θα υποβάλουμε τα συμπεράσματά μας στην Επιτροπή σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα έρθουμε σε επαφή με Ισπανικές Αρχές. Μάλιστα, όλοι οι συναδελφοί μου βρίσκονται σήμερα στην Μαδρίτη, συνομιλούν δηλαδή με τις Ισπανικές Αρχές αυτή τη στιγμή. Θα επανεξετάσουμε λοιπόν τους ισχυρισμούς αυτούς, τους νέους αυτούς ε, ισχυρισμούς και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Ρώσα, βιάζεσαι. Σου δίνω το λόγο πρώτη. Κυρία Σταράς, ευχαριστώ πολύ για του αναφέροντες και ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να ε, εγκαταλείψω την αίθουσα ε, πριν ολοκληρωθεί η εξέταση τη αναφορά. Έχω μια άλλη υποχρέωση. Ε, ακούσαμε την Κομισιόν, η οποία είναι σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο θα ήθελα να κρατήσουμε την αφορά ανοιχτή. Εγώ μίλησα με το Υπουργείο πριν από τη σημερινή συνάντηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης μου είπε ε, ότι ε, είναι δεσμευμένοι και τηρούν την δέσμευση υπογειοποίησης του ε, τρένου ταχύτητας. Ε, θα γίνει μια προσινή παράκαμψη, αλλά τελικά ε, θα, η υπογειοποίηση θα γίνει σε όλο το μήκος το οποίο έχει προβλεφθεί. Πιστεύω ότι αυτό που κάνατε εσείς, ο δικός σας αγώνας, έχει επηρεάσει το Υπουργείο. Μίλησα την περασμένη εβδομάδα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ε, μου επιβεβαίωσαν αυτή τη δέσμευση ότι θα γίνει πλήρης υπογειοποίηση. Όμως, μέχρι ότου γίνει αυτό, κάποιες, ε, για κάποιο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να γίνουν ε, παρακάμψεις. νομίζω ότι έχει συστηθεί ένα συμβούλιο της Κοινωνικής Επιτροπής για την υπογειοποίηση του, τετρών ψηλής ταχύτητας στη Μούρθια. Συμμετέχουν τα συνδικάτα, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι κλπ. Έχει συνέλθει δύο φορές αυτό το, συνέδριο, ε, αυτό το συμβούλιο, αυτή η επιτροπή και νομίζω ότι θα χρησιμεύσει έτσι ώστε να παρακολουθούμε από κοντά τα έργα. Ε, οι, μου λένε ότι η εκτίμηση προγραμματικών επιπτώσεων που είχε γίνει το 2002 ε, ε, ισχύει ακόμα. προσπάθησαν τα έργα να γίνουν σε διαφορετικές φάσεις λόγω της κρίσης, ανάλογα με τα χρήματα που είχαν. Αυτό που μου λένε είναι ότι στις 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε η φάση, το, το κομμάτι Σαντιάγο Δελμαγιόρ, για την υπογειοποίηση ενός τμήματος. Ε, όπως σας είπα θα έχουμε κάποιες προσωρινές ε, ε, παρακάμψεις. Ε, σύντομα θα ξεκινήσει και η φάση της υπογειοποίησης στον, ε, στον τερματικό σταθμό. εγώ σέβομαι και πιστεύω τον Υπουργό Χαίρομαι που δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή Κοινωνικής Διαβούλευσης. Ε, η Κομισιόν έτσι και αλλιώς βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ε, τοπική κυβέρνηση Μούρθια και με το Ισπανικό κράτος, οπότε ας κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου η ίδια η Κομισιόν να μας πει να μας αναφέρει τα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει ε, πιστεύω ότι η αναφορά σας θα ικανοποιηθεί. Thank you very Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους αναφέροντες που είναι εδώ σήμερα. Είναι μακριά η ιστορία αυτή. Ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα η συζήτηση για αυτό το έργο στην Ισπανία και ε, μάλιστα ε, για ένα τρένο το οποίο θα φτάνει υπογείως στη Μούρθια. Ε, η ιδέα ήταν η άφηξη αυτού του υπογείου τρένου και έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμα. Μετά διαπιστώθηκε ότι όταν έπρεπε να ξεκινήσει δεν αρκούσαν τα χρήματα για να γίνει υπόγεια η κατασκευή και η κυβέρνηση τότε είπε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο. Πέραν των όσων συνέβασαν έκτοτε και το τι αλλαγές έγιναν, αυτό το οποίο με ανησυχεί κυρίως αν και με καθησυχάζει λίγο αυτό που είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάποια στιγμή ε, και βάσει ε, εκεί θα έπρεπε να γίνει η κατασκευή σε ε, μια οδό η οποία υπήρχε ήδη. Δεν θα δημιουργούνταν ένα νέο δίκτυο σιδηροδρομικό, αλλά υπήρχε ήδη η γραμμή και ε, από εκεί και πέρα υπήρχε και μία θετική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά οι πολίτες και πάρα πολλοί ε, αρχές λένε ότι άλλαξαν τα πράγματα και αλλάζει συνεχώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων πρέπει ε, λοιπόν να εμπιστευτεί αυτό που τις λένε οι Ισπανικές αρχές. Αν υπάρχουν όμως τόσες πληροφορίες θα πρέπει να μεταβείτε επιτόπου ε, κατά την άποψή μου και να πάτε να δείτε αν όντως έχουν αρχίσει τα έργα. όπως λέει ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι γι' αυτό, θα υπάρξει νέα ε, κοινοποίηση προς τους αναφέροντες και ε, θα δούμε κατά πόσον πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές. Σίγουρα πρέπει να έρθει σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές και μάλιστα ε, αν πάτε στη Μαδρίτη σίγουρα θα πρέπει να πάτε και μέχρι τη Μούρθια για να δείτε οι δύο αν υπάρχουν συντρέχουν λόγοι για να έρθετε σε επαφή ε, και να απαντήσετε και στους αναφέροντες. Ε, να δούμε όλα αυτά τα επιχειρήματα και τα έγγραφα τα οποία αιτιολογούν που λέτε ότι σας ε, προσκόμισε η Ισπανική κυβέρνηση για να διαπιστώσετε ότι όντως όλα πηγαίνουν κατευχήν εγώ εξ ονόματο των φιλελευθέρων πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά σίγουρα μέχρι να επιληθεί το ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να, να εξετάσει επιτόπου το θέμα και να λάβει τις κατάλληλες εγγυήσεις και ότι το αρχικό ε, πρόγραμμα, ε, σχέδιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί αυτό έχει και τη θετική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλιώ να ξεκινήσει ε, διαδικασία επιπαραβάση για το συγκεκριμένο έργο. Ευχαριστώ πολύ. η κυρία Αλμπιόλ. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω τους αναφέροντες και να υπογραμμίσω ότι εδώ και 73 μέρες ε, έχουμε κινητοποιήσει ε, των γειτόνων ε, του τοπικού πληθυσμού που έχουν βγει στους δρόμους ζητώντας να μην χωριστεί στα δύο υπόλοιπους από το τρένο. Ε, φανταστείτε τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες, πώς θα διασχίζουν τις γραμμές από υπόγειες διαβάσεις κλπ. Δύο θέματα θέλω να υπογραμμίσω. Πρώτον, το σχέδιο αυτό έχει αλλάξει. Το τρένο υψηλή ταχύτητα θα φτάσει στη Μούρθια υπέργειο, όχι υπόγειο. Το δεύτερο θέμα που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία έγινε επί ενός σχεδίου το οποίο έχει αλλάξει. Συνεπώς είναι κατακαιρματισμένη, μη επίκαιρη και ανεπαρκής. Ε, λέω κατακαιρματισμένη γιατί το έργο αυτό κατακαιρματίστηκε, χωρίστηκε σε μικρά τμήματα για να αποφευχθεί μια συνολική εκτίμηση περιβαλλοντικής επιπτώσης ε, και ανεπαρκή λέω ε, διότι δεν, η, μελέτη που υπάρχει δεν αφορά το σχέδιο το οποίο υλοποιείται. Συνεπώ και η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ανεπαρκή. Άρα λοιπόν ε, δεν την χάνει σεβασμού η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Τι οποίε είναι θεματοφύλακα η Κομισιόν. Το έχουμε δει και άλλε φορέ αυτό. Σε έργα μεγάλων υποδομών στην Ισπανία, ε, σε ε, πολεοδομικές περιπτώσεις και υποθέσεις Πολύ συχνά αλλάζουν τα σχέδια χωρίς να αλλάζει, χωρίς να επικαιροποιείται η μελέτη περιοριστικών επιπτώσεων κλπ. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή κάνει και πρέπει να κάνει την εξέταση του κατά πόσον είναι επαρκής η παλιά μελέτη, όχι κλπ. Ε, και αν υποδειχθεί ότι χρειάζεται να επικαιροποιηθεί θα πρέπει να παραλύσουν τα έργα. Δεύτερον, περιμένοντας και την απάντηση της Κομισιόν, εμείς θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών της Ισπανίας για να τους εκφράσουμε την ανησυχία μας για αυτό το, αυτή την μπάρα η οποία θα χωρίσει την, ε, ε, για αυτό το φράγμα μάλλον θα χωρίσει την πόλη στα δύο. Ευχαριστώ κύριος Μαρσελέση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες ε, οι οποίοι ήρθαν μέχρι τις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν αυτή την αναφορά. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να ζει κάποιο σε μια πόλη ε, η οποία χωρίζεται από σιδηροδρομικές ε, ράγες. Ε, εγώ πήγα επιτόπου στη Μούρθια και αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 ε, πολίτες στο νότιο τμήμα της πόλης που είναι απομονωμένοι από το κέντρο της πόλης και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες ε, διότι υπάρχει απλώς μόνο μία υπόγεια διάβαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει να ζει κάποιος αυτή την κατάσταση και έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες. Ε, πράγματι, η Ισπανική κυβέρνηση απάντησε ότι δεν άλλαξε η εκτίμηση περιβαλλοντικών υποπτέσεων ε, από το 2012, αλλά αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι πέραν αυτού υπάρχει και ένα άλλο έργο, ε, το οποίο θα κατασκευάσει σε 2-3-4 χρόνια, όσο θα διαρκεί το έργο, μια παράλληλη οδό, η οποία θα είναι υπέργεια. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών υποπτέσεων του 2009. Πολύ καλά λοιπόν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθυνθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων για να δει τι γίνεται με αυτή την παράλληλη οδό η οποία υποτίθεται ότι θα λειτουργεί όσο καιρό θα είναι να εξελίξει τα έργα. Διότι αν έχουμε έργα για κάποια χρόνια ε, και ε, ταυτόχρονα έχουμε και μια παράλληλο εδώ, πρέπει να δούμε και όλες τις συνέπειες που θα υπάρχουν. Είναι αρκετές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ουσιαστικά ε, θα αναδιαμορφωθεί η κυκλοφορία στην πόλη, αλλά μπορεί να υπάρχουν και συνέπειες για την υγεία των κατοίκων και θα υπάρχει και συνέπεια για την ε, χλωρίδα της περιοχής. Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ανησυχεί επίσης και αυτό που είπαν οι αναφέροντες ε, για τη σύμβαση του Άρχους. εγώ ε, κατάλαβα ότι πήγανε στον εισαγγελέα αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος και δεν έλαβαν απάντηση και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρωτήσει και την Ισπανική κυβέρνηση για τα όσα συνέβησαν με την ε, εισαγγελία περιβάλλοντος και το κατά πόσον τηρούνται τα της σύμβασης του Άρχους. Ε, αντιλαμβάνομαι πλήρως ε, τους φόβους των αναφερόντων, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που τους δίνονται υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Για παράδειγμα και στο Βαγιαδολέιθ υπήρχε υπόσχεση να υπάρχει υπόγειο ε, και εδώ ε, πλέον έχουν οριστικοθεί τα πράγματα, είναι πλήρες υπέργειο το έργο, δεν υπάρχει τίποτα υπόγειο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ισπανία αυτή τη μορφή. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα σχολιάζουμε εδώ στην Επιτροπή των Αναφορών. Θα θυμάστε για παράδειγμα ότι είχαμε και ε, άλλα αντίστοιχα περιστατικά της Ισπανίας σε θέματα χωροταξίας ε, και υποστηρίζω και την πρόταση της ε, συναδέλφου να πάτε επιτόπου μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί ουσιαστικά δημιουργείται ένα φυσικό φράγμα στην πόλη που χωρίζει χιλιάδες πολίτες. Υποστηρίζω λοιπόν και εγώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά μέχρι να υπάρχει σαφή σαφής σωστή ε, του έργου από την ε, Ισπανία. Ευχαριστώ κυρία Βαλίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες για τον αγώνα τους. Και όπως είπε ο συνάδελφος μόλις τώρα, η τάση σε αυτή την ε, επιτροπή είναι και το βλέπουμε συχνά με την κεντρική κυβέρνηση και με τις περιφερειακές κυβερνήσεις στην Ισπανία ε, να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη τακτική ε, της, του κατακαιρματισμού των μεγάλων έργων σε μικρότερα προκειμένου να αποφευθεί μια συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι ένα τρίκ που κάνουν ε, έτσι ώστε να προχωρήσουν με έργα τα οποία αλλιώς δεν θα γινόντουσαν δεκτά και η Κομισιόν θα πρέπει να αρχίσει να το αντιλαμβάνεται και να κάνει κάτι, διότι είναι μια πρακτική η οποία γενικεύεται ε, τελευταία στην Ισπανία. Όπως έλεγε και η Φλωρένσα, το είδα, ο, όπως το είπε ο Φλόρενς, ε, το είδαμε με το πάρκο της Δονιάνα και το είδαμε και με άλλα, το βλέπουμε και πολλά άλλα έργα. Ε, Νομίζε η κυβέρνηση ότι ε, με την ε, υπογειοποίηση ενός μικρού τμήματος ε, λύνονται όλα τα προβλήματα. Η Κομισιόν δεν πρέπει να το δεχτεί αυτό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα του, της απομόνωσης συγκεκριμένων γειτονιών. Υπάρχουν προβλήματα με τις ακουστικές μελέτες κλπ. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα της πρόσβασης στην πληροφόρηση εκ μέρους των πολιτών τα δικαιώματά τους ε, παραβιάζονται και η Κομισιόν κάτι πρέπει να κάνει. Στην τελευταία διαδήλωση πάνω 50.000 άτομα βγήκαν στο δρόμο υπέρ της υπογειοποίησης και η απάντηση ποια ήταν, ήταν τα γκλόπ των αστυνομικών. Σε ανθρώπους που απλώς ε, διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Έτσι απαντάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να αντιληφθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και η, και τοπική κυβέρνηση της Μούρθια ότι το έργο αυτό δεν το θέλουμε αυτόν τον τρόπο. Ε, ε δεν το θέλει με αυτόν τον τρόπο ο τοπικό πληθυσμό. Ο Υπουργό, από την άλλη μεριά, όπω είπε η κυρία Σταρά, μπορεί να είπε κάποια πράγματα και να υπόσχεται υπογειοποίηση, αλλά εγώ θυμάμαι τις, τι είχε πει ο Υπουργό ε, ω ε, δήμαρχο Σανταντέρ. Ε, τι είχε πει ω δήμαρχος του Σανταντέρ για, την, ε, για τα πορίσματα της έρευνα για το, ε, τρε, για το τύχημα, τύχημα της Άβυλα ε, και θυμάμαι ότι όταν έγινε υπουργό τα έκανε γαργάρα. Ελπίζω λοιπόν να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Παρακαλώ η Κομισιόν να επισκεφθεί επιτόπου τα έργα. Άλλη είναι η κατάσταση επιτόπου και άλλη στα γραφεία σας και να το ξανασυζητήσουμε όταν έχουμε στα χέρια μας όλες τις, όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η Soledad. Καλώς και πάλι στην Επιτροπή. Ε, έχω πολύ καιρό να σας δω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Καμπεθόνο Ρουίθ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους αναφέροντες και νομίζω ότι η φωτογραφία αυτής της ε, τόσο πολυπληθούς ε, ε, διαδήλωσης δείχνει τι νιώθει ο κόσμος της Μούρθια. Και χαίρομαι που σήμερα αιτιολογήθηκαν τα πράγματα και νομίζω ότι αιτιολογήθηκε το γεγονός ότι τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα με διπλό τρόπο και από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το έργο και το πώς φτάσαμε εδώ ουσιαστικά ε, η πόλη ξέρει πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να φτάσει το τρένο στην πόλη της ε, και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι ηθήνοντες, οι οποίοι είναι ερμόδιοι αυτή τη στιγμή, αλλά και όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι ορισμένες φορές κάνουμε πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι οι πολίτες της Μούρθια μας λένε σαφώς ότι δεν πρέπει να γίνονται έτσι τα πράγματα. Ε, γιατί μου ήρθε ένα διαφυσβήτητο ότι πρέπει να είναι υπόγειο το έργο και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την προπόθεση και από εκεί και πέρα να αναζητήσουμε τις λύσεις που πρέπει να προτείνουμε. Στην Ισπανία έγινε μια πολύ σημαντική επένδυση ε, για τις υποδομές για αυτά τα τρένο υψηλής ταχύτητες ε, σε μεγάλες περιοχές της επικράτειας, αλλά υπάρχουν κάποιες περιοχές, κυρίως ε, ε, τις πιο απομακρυσμένες, που δεν έχει φτάσει ακόμα το τρένο και ε, δεν φαίνεται να είμαστε ακόμα τόσο αποτελεσματικοί ή να έχουμε τη βούληση για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Η Μούρθια είναι περιοχή της νοτιοανατολικής Ισπανίας και πρέπει και αυτή να είναι διασυνδεδεμένη, να είναι καλά συνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ισπανία και με άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Ισπανίας και νομίζω ότι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και για τη Μούρθια και για τους πολίτες. Πρέπει να υλοποιηθεί το έργο, αλλά με τις προϋποθέσεις που επιθυμούν, γιατί είναι οι μόνες που είναι κατάλληλες για μία πόλη η οποία δεν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα να κοπεί στα δύο. Ε, διότι δεν μπορεί επειδή ε, θα φτάσει ένα τρένο να κοπεί η πόλη στα δύο. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει το θέμα, διότι ακούγοντας ε, ε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν έχει τηρήσει τα υπεσχημένα η Ισπανική κυβέρνηση και πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσει ε, πισταμένα το έργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα φτάσετε σε κυρώσεις, δεν με ενδιαφέρει το, ότι, το αν θα υπάρξουν κυρώσεις ή όχι. Πρέπει η Μούρθια να έχει το τρένο της υπόγειο. Και θα πρέπει να μας πείτε και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης με τις Ισπανικές Αρχές, οι οποίες όπως μας λέτε, είναι σε επαφή μαζί σας και αν έγινε αυτή η απαραίτητη αλλαγή του έργου ε, και αν έχει αλλάξει και στάση κυβέρνηση. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν ε, να είστε σε επαφή με την Επιτροπή Αναφυρών για να βλέπουν και αναφέροντα ότι είμαστε χρήσιμοι, ότι εισακούστηκε το αίτημά τους και θα βρεθεί η λύση που αναζητούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now it's time. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξαναδώσω το λόγο στους αναφέροντες. Oh, sorry. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, είναι καπριτσιό το γεγονό ότι βρισκόμαστε εδώ τόσοι από τόσα διαφορετικά κόμματα. Γνωρίζουμε πώς, γίνεται, πώς ασκείται η πολιτική στην Ισπανία και οι κάτοικοι της Μούρθια χρησιμοποιούν το ένα εργαλείο που έχουμε έτσι ώστε τα λόγια να γίνουν πράξη. Ε, οι, οι λέξεις ε, δεν ε, θα πρέπει να παραπλανούν την κοινή γνώμη. Χρειάζεται να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και η Κομισιόν, εκτός από αυτά που μας είπε ότι θα κάνει στην, στις επαφές της και ενημερωτικά θα πρέπει να επισκεφθεί την ε, περιοχή διότι εκεί θα δει μια πληγή μέσα στην ίδια την πόλη. Εμείς τη βλέπουμε εδώ και χρόνια. Αυτά που λένε οι γείτονες εκεί είναι πραγματικά, είναι η πραγματική κατάσταση. Αφενός παραβιάζονται οδηγίες και η νομοθεσία, ε, παρακάμπτοντας ε, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και δεύτερον ε, η κατάσταση ε, ε, για αυτούς είναι πραγματικά πολύ άσχημη. Σκεφτείτε ποια θα, τι θα υποφέρουν τα, αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι, αυτά τα φτυχά, φτωχά προάστια που βλέπουν να διαχωρίζονται από το κέντρο της πόλης. Ε, και δεν μας τα είπαν όλα γιατί είναι άνθρωποι ταπεινοί, διακριτικοί ε, αλλά πραγματικά υποφέρουν πολύ και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Η Κομισιόν θα πρέπει να τους εγγυηθεί όλα τα δικαιώματά τους. Είναι πολίτες οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν να βελτιώσουν την ε, σύνδεσή τους με την υπόλοιπη πόλη. Θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε και να τους συνοδεύσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να υλοποιηθεί η υπογειοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα Σέντερ, καλώς ήρθατε. Ζητώ συγγνώμη, βρισκόμουν σε μια άλλη συνεδρίαση που ασχολείται με θέματα ενέργειας για τη Μεσόγειο, είμαι μακριά. ορίζω τους ε, αναφέροντες. Ε, συναντήθηκα μαζί τους Άκουσα τα παραπονά τους και τις διεκδικήσεις τους, τα αιτήματά τους. Είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Έχουν γίνει αλλαγές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την αναφορά τους ε, κατάφεραν πραγματικά να κινήσουν τα γρανάζια ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. με δημόσια έργα που αφορούν ε, υποδομές ε, μεγάλες όπως αυτό το τρένο ψηλής ταχύτητας αλλά και άλλου τύπου υποδομές. Θα το δούμε αυτό και στους ευρωμεσιακούς ε, διαδρόμους και τα δίκτυα μεταφορών. Με τέτοιου είδους έργα λοιπόν χρειάζονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, οι οποίες θα βασίζονται και σε διαβούλευση με, το, με τους πολίτες με στόχο να γίνει πιο να γίνουν πιο ήπιες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτά τα έργα. Και αυτό θα πρέπει να δούμε και στη Μούρθια. Το πώς η υλοποίηση αυτής της ε, ε, υποδομής, αυτών των υποδομών, επηρεάζει την καθημερινή ζωή και το περιβάλλον στην Μούρθια. Η απόφαση για την υπογειοποίηση ε, είναι πολύ σημαντική Με την Καταλωνία και την Τζιρόνα ε, ε, η αντίστοιχη υπογειοποίηση αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα αποφύγουμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει σωστά και θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει για να τις αντιμετωπίσουμε αυτό το ερώτημα. Την περασμένη εβδομάδα ο υπουργό ήταν στο Στρασβούργο και μιλήσαμε για αυτό το θέμα σε μια συνάντηση που είχα μαζί του. Και εδώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ τους αναφέροντες γιατί πραγματικά οι κινητοποίησεις τους δίνουν αποτέλεσμα. Μπορεί να μην είναι αρκετό αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα ε, ή να μην είναι έγκαιρο όσο θα το θέλαμε. Παρόλα αυτά το Υπουργείο έχει ευαισθητοποιηθεί και πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός. Συνεπώς να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά έτσι ώστε στις διαβουλεύσεις της Κομισιόν να ε, εξετάσει το θέμα και να μας απαντήσει γραπτός έτσι ώστε να δούμε ακριβώς που βρίσκεται το θέμα. Έτσι ώστε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να πάρουμε μια δεύτερη απόφαση. Σας βεβαιώ ότι ο αγώνας σας, οι κινητοποίησεις σας άλλαξαν την κατάσταση σε ευρωπαϊκό πέδο και ελπίζω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης της Ισπανίας. Ας διατηρήσουμε την πίεση όμως, όπως είπε και η Πρόεδρος, να ζητήσουμε από την Κομισιό να έρθει σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές, να πάρει από, απαντήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης ε, και να παρακολουθήσουμε την υπόθεση στενά. Ευχαριστώ και τώρα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους αναφέροντες ε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Έχετε δύο λεπτά. Έγιναν κάποιες αναφορές ε, στην ανάγκη υπογειοποίησης και στην άφηξη του τρένου. Κανείς ε, δεν το αμφισβητεί αυτό. Μην θεωρήσει κανείς ότι δεν θέλουμε να φτάσει το τρένο υψηλή ταχύτητα στη Μούρθια σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλουμε να είναι συμβατά τα δύο πράγματα και είναι προτεραιότητα να είναι υπόγειο ε, το τρένο το οποίο θα φτάσει. Εδώ και 30 χρόνια δίναμε τη μάχη και τότε δεν υπήρχε στον ορίζοντα το θέμα του τρένου το θέμα ήταν αν θα υπάρχει υπόγεια ε, οδός με τρένο ή χωρίς. Ε, και ήρθε και το τρένο, εμείς σε καμία περίπτωση δεν είμαστε κατά, αλλά πρέπει να είναι υπόγειο όπως συμφωνήθηκε το 2006. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε να έχουμε ένα υπέργειο τρένο και μάλιστα ε, χωρίς κανένα νόημα ε, και υποχρεωτικά, διότι το ε, τρένο το οποίο θα είναι υπέργειο θα χωρίσει και θα διαταράξει τις υπάρχουσες γραμμές. Ε, έχει τελείως διαφορετικές περιβαλλοντικές συνέπειες για την ηλεκτρική γραμμή, με πλήρη ε, ε, προστασία και θα υπάρχει ένα τείχος το οποίο θα χωρίσει την πόλη στα δύο οριστικά. Και υπάρχει και τεκμηρίωση την οποία θα μπορούσα να σας προσκομίσω. Έγιναν ε, απόπειρες να παραλύσει ένα σχέδιο το 2011 υπήρχε ένα έργο το οποίο σταμάτησε το 2012, αλλά ταυτόχρονα έγινε κάτι αντίστοιχο το 2013 και το 2014. Έχω μπροστά μου τα σχετικά έγγραφα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε και κατακυρώθηκε και σε κάποια επιχείρηση. Ε, μετά από ένα χρόνο αποσύρθηκε η πρόταση για την επιλογή του νέου έργου το Νοέμβριο του 2014. Αυτό το πήγε νέλα, το ναι ή όχι, το ξεκινάμε και μετά σταματάμε, ε, υποψίασε τους ε, και θεωρήσαμε ότι δεν είναι σοβαρή η πρόταση και αν ε, γίνει υπέργειο στην επιφάνεια το έργο θα παραλύσει το έργο της υπόγειας ε, οδού που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Αν αρχίσατε τη δουλειά σας πάνω στο θέμα αυτό πριν 30 χρόνια, νομίζω ότι θα έχετε καταφέρει να ε, επιστήσετε την προσοχή πολλών ε, στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε για τον αγώνα σας και το πάθος σας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε το θέμα αυτό κρατώντας ανοιχτή την αναφορά, να στείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, επισημένοντας τα εξής. Πρώτον, έλλειψη επικαιροποιημένης ε, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης να ρωτήσουμε σχετικά με την συμμόρφωση ή μη με τη σύμβαση του όρχους, όπως ανέφερε συνάδελφος. Και τέλος, ε, θέλουμε απόλυτη δέσμευση ότι υπογείως ε, θα πραγματοποιηθεί το έργο αυτό και αποκλειστικά υπογείως. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε και ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω βρισκείστε σε συνεχή διάλογο. Παρακαλώ λοιπόν να ενημερώσετε και εμάς σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου σας με τις Ισπανικές Αρχές. Αυτά μπορούμε να κάνουμε νομίζω. Θα μπορούσαμε φυσικά επίσης να στείλουμε το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών προς ενημέρωση. Αυτά νομίζω μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνείτε? Όλοι γνέφουν καταφατικά και να επισημάνω στους ε, αναφέροντας ότι δεν είναι πάντα εύκολο να προεδρεύει κανείς ε, στην Επιτροπή μας, ε, αλλά στην περίπτωση αυτή όπου οι συνάδελφοι από όλε τις πολιτικές ομάδες συμφωνούν είναι μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε, σας ευχαριστούμε που ασχολείστε με το θέμα αυτό που αφορά την περιοχή της Μούρθια, μια τόσο ωραία περιοχή της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ε, παρακαλέσω να αποχωρήσετε ήσυχα και γρήγορα από την αίθουσα, διότι έχουμε και άλλες αναφορές να συζητήσουμε. Ε, θα ήταν πολύ καλύτερο αν μπορούσατε να τις συζητήσετε εκτός της αιθούσης. Can I ask my colleague, Mrs. Παρακαλώ, η συνάδελφος κυρία Αλμπιόλ. Can I ask Mrs. Albiol to escort the petition? Παρακαλώ η κυρία Αλμπιόλ να συνοδεύσει τους ε, αναφέροντες ε, κατά την αποχώρησή τους από την αίθουσα και να συνεχίσετε τη συζήτησή σας εκτός της αιθούσης. Mrs. Albiol. Κυρία Αλμπιόλ, παρακαλώ. Can I ask you kindly to escort the, the petitioners outside the room so that we can continue? Μπορείτε παρακαλώ να συνοδεύσετε τους αναφέροντες ε, και να συνεχίσετε τη συζήτησή σας μαζί τους εκτός της αιθούσης. Now it's high time to turn to the Danish petition. Να προχωρήσουμε τώρα στην δανέζικη αναφορά. σχετικά με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη Δανία για την επέκταση της υδατοκαλλιέργειας. Πρόκειται για την αναφορά 578. Είναι παρούσα η Εύα Μαρία Βίνια Χασπίλε. Ε, αναφέρουσα και έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη σημαντική αυτή υπόθεση που έχει να κάνει με την παραβίαση από πλευρά της Δανέζικης νομοθεσίας αρκετών νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικά με τα ύδατα. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας διάφορους πολιτικούς και πολίτες από την Δανία που δεν μπορούν να είναι παρόντες διότι μόλις είχαμε ε, δημοτικές εκλογές ε, στην Δανία. Το θέμα αυτό ε, έχει να κάνει με την πρόθεση της κυβέρνησης της Δανίας να επιτρέψει την αύξηση της ρήπανσης στο Κάτεγκατ και τη Βαλτική με τον ε, νόμο υπαριθμών 111 ε, επιτρέπεται περισσότερη ρήπανση από νητρικά και φωσφορικά άλατα και την γενική επιδείνωση του ε, θαλάσσιου περιβάλλοντος με ευτροφισμό εις βάρος της βιοπικιλότητας, επίσης θέματα που σχετίζονται με τα ειζήματα και χωροκατακτικά είδη. Ε, θα ήθελα να σας αναφέρω λοιπόν καταρχάς το θέμα της ρήπανσης, ε, δεύτερον τις αντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τρίτον ε, την σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η οδηγία για τα ύδατα λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί η θα πρέπει να μειωθεί η παρουσία ουσιών που οδηγούν στον ευτροφισμό. Ε, αυτή τη στιγμή το 95% των παράκτιων υδάτων της Δανίας δεν συμμορφούνται με αυτό. Παρ' όλα αυτά η Δανία πιστεύει ότι ε, έχει δημιουργηθεί ε, περιβαλλοντικό περιθώριο, διότι η Δανία έχει μειώσει κάποιες άλλες τιμές. Αλλά αυτό δεν υπάρχει, αυτός ο όρος δεν υπάρχει ούτε στην επιστήμη ούτε στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις ηχθειοκαλλιέργειας να ρηπαίνουν ε, με 800 ε, επιπλέον τόνους νητρικών και 96 επιπλέον τόνους φωσφορικών αλάτων. Ε, και ο νόμος αυτός προβλέπει αντιστάθμισμα για παράδειγμα, εάν φιλτράρει κανείς το πλανκτόν, μπορεί να έχει περισσότερο περιθώριο ε, να ε, ρηπαίνει. Και το αποτέλεσμα της ε, καλλιέργειας μυδιών όσον αφορά την απορρόφηση νητρικών αλάτων δεν έχει αποδειχθεί. Επιπλέον, τα μαλάκια εξαντλούν το οξυγόνο και αφήνουν πίσω Άλλε ουσίε όπω είναι τα αντιβιωτικά και αντιρρυπαντικές ουσίε. Η αντιστάθμιση δηλαδή με ε, αυτή τη μέθοδο δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. Ανησυχούμε σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον στο κάτε-κάτε και ε, στο Τζούσλαντ καθώ επίσης και στι γειτονικέ χώρες, κάτι που δεν έχει ληφθεί υπόψη. Η εξάντληση του οξυγόνου ε, θα είναι καταστροφική για το θαλάσσιο περιβάλλον ε, καθώ και για τον τουρισμό, διότι κανείς δεν θέλει να βλέπει ψόφια ψάρια. Επίσης, ε, χρησιμοποιείται χαλκός στους κλοβούς και αποτελούν επιπλέον ζημιά για το περιβάλλον. Επίσης, δεν υπάρχει περιβαλλοντικό περιθώριο για τη χρήση φαρμάκων ε, στις εγκαταστάσεις ηχθειοκαλλιέργειας ε, και ε, τα χωροκτακτικά είδη που χρησιμοποιούνται στην ηχθειοκαλλιέργεια θα είναι επίσης πολύ βλαβερά για την βιοπικιλότητα. Ε, ο νόμος 111 ε, επιτρέπει η αντιστάθμιση της ε, ρήπανσης με χρήση μεταξύ άλλων καλλιέργειας μηδιών. Αυτό δεν αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο ε, αυτό που αντίκειται στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι το να ε, θεωρείται ότι μία πιο καθαρή περιοχή μπορεί να αντισταθμίσει άλλες εντός των εθνικών ποσοστώσεων. Η οδηγία, για την... η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα σημειώνει ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε περισσότερη ρήπανση και θα πρέπει να πραγματοποιείται ε, ε, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν ε, οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα που θα δείξει ότι όχι μόνο θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, αλλά ότι θα υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη λόγω του τουρισμού. Ε, συμπερασματικά, ο νόμος αυτός αντίκειται στις αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα Ήδατα και της οδηγίας πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική. Υπάρχει εναλλακτική λύση, τα χερσαία συστήματα ηχθειοκαλλιέργειας που ανακυκλώνουν το νερό με ανακυκλοφορία ύδατος ε, και έχουμε ε, Μάλλον ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, φροντίσουν για την εφαρμογή των οδηγιών αυτών στη Δανία για να σταματήσει η εγκατάσταση νέων η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ηχθή καλλιέργεια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ δουλειά έχετε σήμερα το πρωί, σα ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όταν έρχομαι, μου αρέσει να, ε, ε, να εξετάζω ταυτόχρονα διάφορε υποθέσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το, η ρήπανση από νητρικά είναι σημαντικό πρόβλημα σε όλη την βορειοδυτική Ευρώπη, αν όχι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δραστηριοποιηθεί πολύ στο θέμα αυτό. Είχαμε διάφορες δικαστικές υποθέσεις ε, κατά διαφόρων κρατών μελών. Ε, σίγουρα δεν έχουμε φυσικάσει στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που έχουμε σήμερα, τα μέτρα αυτά αποτελούν ε, μέτρο της ε, δέσμης, ε, μέρος της δέσμης μέτρων της Δανίας για τα τρόφιμα και την γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν καταρχάς να εξεταστεί η νομιμότητα των, των θέματων αυτών. Και την 1η Ιουνίου 2017 υπάρχει η τροπολογία ε, για την νομική πράξη αυτή. Αποτελεί όμως εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό, όπως περιέγραψε και η αναφέρουσα. Έτσι λοιπόν υπάρχει νομική βάση για τον Υπουργό να υιοθετήσει περαιτέρω κανόνες. Ε, η εξουδιώτηση αυτή δεν αποτελεί από μόνη της σε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, και με βάση τα ε, στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα ο Υπουργός αυτή τη δυνατότητα. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας, τα μέτρα που έχει λάβει η Δανία στη συγκεκριμένη υπόθεση, που έχουν να κάνουν δηλαδή με τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν δείχνουν να υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι σχετικές δυνατότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρκρετ Άουκεν. Θα μιλήσω δανέζικα ε, σήμερα, διότι ξέρω ότι υπάρχουν ε, διάφοροι στη Δανία που παρακολουθούν την υπόθεση. Αλλά και στον Πίτερ και στην Σεσίλια θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα που αφορά και τη Γερμανία και τη Σουηδία. Και ακούσαμε και από τις βαλτικές χώρες ότι γνωρίζουν ότι η Δανία στο θέμα αυτό έχει ενεργήσει σαν ε, να είναι τελείως απομονωμένη. Ε, δεν ε, έχει ενημερώσει όσους θα έπρεπε και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχετε πει ότι... Γιατί δεν έχετε ασχοληθεί με το γεγονός ότι η θαλάσσια στρατηγική θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με τον ίδιο τρόπο με την Helcom, διότι η θαλάσσια στρατηγική είναι σχετικά νέα, αλλά την χειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο με την Helcom, ε, αλλά η ε, Δανία ενεργεί σαν να είναι μόνη της. Ε, είπανε ωραία όσον αφορά τη θαλάσσια στρατηγική, ενεργήσαμε πιο γρήγορα σε κάποια πράγματα και γι' αυτό μπορούμε να αντισταθμίσουμε με περισσότερη ρήπανση. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και κάτι ακόμα που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η Δανία μέχρι την κυβέρνηση αυτή είχε ε, αντιμετώπιζε συνδυασμένα την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και αυτήν για τη θαλάσσια στρατηγική. Δεν θεωρούσε ότι ε, τα ύδατα σταματάνε στα σύνορα. Αλλά τώρα πια έχει διαχωρίσει τις ε, δύο αυτές ε, οδηγίες, διότι είχαμε κάποιες καταδίκες σε σχέση με την οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική που δείχνουν ότι η Δανία δεν έχει εκπληρώσει καθόλου τις υποχρεώσεις της. Έγιναν κάποιες ε, δοκιμές όσον αφορά την καλλιέργεια μυδιών ε, σε ένα φιόρντ της Δανίας, ε, όπου υπήρχαν καλά αποτελέσματα, αλλά εκεί ήταν φιόρντ, ενώ εδώ μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα. Και η συγκεκριμένη ακτή θα επηρεάσει και τη Σουηδία, διότι έχουμε εκεί τον δυτικό ανεμό στα βόρεια, που κινεί τα πράγματα προς τα ανατολικά, στη Σουηδία δηλαδή. και η Βόρεια Γερμανία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορείτε επιτέλους μία φορά να ενεργήσετε προτού πάνε τα πράγματα στραβά. Μας λέτε ότι αφού δεν έχει πάει τίποτα στραβά, αφού ο υπουργό δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα αυτή την εξουσιοδότηση, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτή είναι η στρατηγική ε, της αυτοψίας. και οι αναφέροντες μου είπαν ότι αυτή τη φορά έχουμε ένα νόμο που έχει θεσπιστεί, ενώ άλλες φορές ε, είχαμε περιπτώσεις ε, νομοσχεδίων που δεν είχαν ε, υιοθετηθεί ακόμα. Και τώρα που έχουμε την νομοθεσία μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε αν δεν πάνε στραβά τα πράγματα. Όχι, να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας και να αντιδράσετε διότι η Δανία ε, έχει αντιδράσει τελείως απομονωμένα και ξέρω ότι οι κακόμοιροι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ δεν ε, ε, είναι στο, στην κορυφή της ιεραρχίας, ούτε ασχολείστε μόνο με το περιβάλλον. Αλλά θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να μην πάνε στραβά τα πράγματα στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάρλσον. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Εδώ και πολύ καιρό παρακολουθώ το θέμα αυτό με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ ανησυχία. Η κυβέρνηση της Δανίας ε, έχει δώσει τη δυνατότητα διεύρυνσης της ηχθυγοκαλλιέργειας ε, στη θάλασσα και ακούμε εδώ ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος λόγω των θρεπτικών ουσιών που εκλείονται. Ε, θα ανατρέψουν την ε, φυσική ισορροπία στις θάλασσες. Και γι' αυτό ήθελα πολύ να ακούσω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι και εγώ περίμενα μια πιο σαφή απάντηση. και περίμενα να ακούσουμε ότι πρόκειται για σαφή παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα τι χρειάζεστε επιτέλους προτού να λάβετε μια σαφή απόφαση. Αυτό μου λείπει εδώ, διότι νομίζω ότι με την ε, ικανότητά μου να αξιολογήσω την κατάσταση και ακούγοντας τους εμπειρογνώμονες μου φαίνεται ότι είναι σαφές ότι έχουμε εδώ παραβίαση της νομοθεσίας. Και όπως λέει η Μαρκρέτα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχει γίνει η ζημιά. Και σήμερα το πρωί μόλις άκουσα από τον Δανέζικο τύπο ότι υπάρχουν νέες αναφορές που δείχνουν ότι η ποσότητα του αζότου στις ε, θάλασσες γύρω από τη Δανία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ κακή ιονή και ελπίζω και επιθυμώ να έχουμε περισσότερη σαφήνεια στο θέμα αυτό. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο πάλι στην αναφέρουσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ την ε, Κομισιόν, ευχαριστώ όλους και όλες σας. Ευχαριστώ πολύ που εξετάζετε την αναφορά μας. Η απάντηση που δόθηκε από τους ευρωβουλευτές ε, ε, δεν είναι πολύ ικανοποιητική. Η απάντηση της Κομισιόν μάλλον δεν είναι ικανοποιητική. Βασίζεται ένα τεχνικό επιχείρημα θα πρέπει να δράσουμε πριν γίνει μόλις των θαλασσών. Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι γνώμες ε, των γειτονικών κρατών. Η Κομισιόν έχει ακούσει ακούσει ποτέ την έννοια του περιβαλλοντικού χώρου που μπορεί να μολυνθεί. Δεν υπάρχει αυτό στην επιστήμη, δεν υπάρχει ως ορολογία. Ε, να τονίσω το τελευταίο που υπόθηκε. Είναι εκπληκτικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πάρει θέση. Αυτό είναι ακριβώς το περιβαλλοντικό περιθώριο που ε, έχει εφεύρει, ο νέος αυτός όρος που έχει εφεύρει η ε, δανέζικη κυβέρνηση. Θα πρέπει τουλάχιστον να επιμείνετε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς ε, να το χρησιμοποιήσει. Και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους εδώ, την Σεσίλια, τον Πίτερ και άλλους, να ευαισθητοποιήσετε και τις δικές σας αρχές ε, απέναντι στο θέμα αυτό, διότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν φαίνεται να ε, έχει θυγεί που η Δανία έχει ενεργήσει τελείως εγωιστικά και εθνικιστικά. Ναι, αλλά από την άλλη, λέει η Πρόεδρος, ε, η νομοθεσία του 2017 της Δανίας δεν είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι δανέζικη νομοθεσία, την οποία ίσως να μην ε, εφαρμόζει η Δανία. Μπορεί να είναι πολύ καλός νόμος, αλλά εάν δεν εφαρμόζεται στην πράξη δεν έχει κανένα νόημα. Η κυρία Όκεν. Όταν μιλάμε για τη Βαλτική, για το Κάτεγκατ μιλάμε για περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Δανία εκεί δεν μπορεί να θεσπίζει δικούς της νόμους. Είναι θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέμα που αφορά τη Σύμβαση Χέλκον Και η Δανία συμπεριφέρεται σαν να πρόκειται για καθαρά εθνική νομοθεσία και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει κάνει μια παρατήρηση ε, αντί απλά να περιμένει να δει αν θα πάνε τα πράγματα στραβά. Πρόεδρος, θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά ενώ θα έπρεπε να είναι σαφές, μου προκαλεί λίγο πονοκέφαλο, διότι έχουμε στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βαλτική, την οποία δεν άκουσα να αναφέρει κανείς μέχρι τώρα και ίσως αυτό θα μπορούσε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική για τη Βαλτική είναι ένα έγγραφο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί και όχι απλά να είναι ένα έγγραφο στη βιβλιοθήκη. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό. Η εθνική νομοθεσία ε, συμμορφούνται πλήρως με τη στρατηγική αυτή και τα μέτρα που αναφέρονται στη στρατηγική έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Δανίας. Αυτό είναι το ένα. Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, θα ζητήσουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ε, και τη στρατηγική της Βαλτικής. Και θα απευθυνθούμε στο Δανέζικο Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα τους εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας ε, στο θέμα αυτό και θα τους συστήσουμε να μην χορηγήσουν άδειες για νέα έργα με βάση το νέο νόμο. Θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα πιο σφαιρικά. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες. Εμένα αυτό με απασχολεί πιο πολύ. Εκτός μικροφώνου η κυρία Όκεν. Και αυτό το περιβαλλοντικό περιθώριο, αυτός ο όρος ε, που αναφέρει η κυβέρνηση της Δανίας. Ε, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημάνει ότι δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρόεδρος, αυτό που βλέπουμε όχι μόνο στη Δανία και δεν ε, θα σας παραθέσω τα λόγια του Σέξπιρ, ε, τα ίδια τα βλέπουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάθε κράτος μέλος ενεργεί εγωιστικά, δεν ασχολείται με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το τι κάνει η Δανία λοιπόν έχει συνέπειε ε, για το σύνολο της Ευρώπης και ιδιαίτερα για την περιοχή της Βαλτικής, ε, για τη Γερμανία, για τη Σουηδία και τι άλλες χώρες εκεί. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα το επισημάνουμε αυτό στην επιστολή και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε ενισχυμένη συνεργασία, να το πούμε έτσι, ε, με εσά στο θέμα αυτό και σας καλούμε να εξετάσετε την στρατηγική για τη Βαλτική την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στη Δανία. Hey, Peter. Ο Πίτερ, ε, κυρία Πρόεδρε, θα με ενδιέφερε και η γνώμη των ε, θεματικών επιτροπών μας. Ε, είναι λοιπόν ένα θέμα κατάλληλο για το δίκτυο ΠΕΤΗ οι ε, Επιτροπές Περιβάλλοντος και Αλίας ε, ε, θεωρούν ότι είναι εντάξει τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει εμάς το θέμα, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και την άποψη των θεματικών επιτροπών Αλίας και Περιβάλλοντος. So we send a letter to... Ωραία, να κάνουμε και αυτό. Να στείλουμε μια επιστολή στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Επιτροπή Αλίας και να ζητήσουμε και από τον υπεύθυνο του τμήματος να το θέσει σε ένα από τα θέματα του Petty Network, του δικτύου της Επιτροπής Αναφορών, διότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με το καλό να επιστρέψετε στη Δανία και περνάμε τώρα στο σημείο 16, 1 και 2. Παρουσίαση της μελέτης του EPRS, ε, της ε, του Κέντρου Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θερινή ώρα και την ε, οδηγία του 2006 αξιολόγηση επιπτώσεων εκ των Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της, ε, του EPRS. Παρακαλώ να σας δώσω το λόγο, η κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας ε, για τη θερινή ώρα. Εργάζομαι για το Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνέταξα αυτή τη μελέτη κατόπιν αιτήματο τη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, ζήτησε να εξετάσουμε τον αντίκτυπο τη θερινή ώρα ε, σε αρκετού τομεί, ε, στην ενέργεια, στην οικονομία και στην υγεία. Μπορείτε να το βρείτε και διαδικτυακά και υπάρχει και ένα μικρό αριθμό ε, εκτυπωμένων αντιγράφων στην είσοδο της αίθουσα. Καταρχάς, θα ήθελα να σας θέσω τη θερινή ώρα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα αναφέρω τον αντίκτυπο της θερινής ώρας σε διάφορους τομείς και επίσης θα εξετάσουμε και την άποψη της κοινή γνώμης πριν ε, καταλήξουμε σε κάποιες ε, σκέψεις για πιθανές εναλλακτικέ λύσεις η ιδέα της θερινής ώρας είναι να εκμεταλλευτούμε το φως της ημέρας. Γι' αυτό ακριβώς ε, και την αποκαλούμε ημέρα εξοικονόμησης, υπάρχουν και τα αρχικά VST. Ε, μετά από την ισομερία, την άνοιξη, αλλάζουμε την ώρα, πηγαίνει μια ώρα μπροστά και στο τέλος Οκτωβρίου ε, γυρίζουμε και πάλι στην ε, ώρα. Εκφύσεως η θερινή ώρα αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητιέται συχνά ιδιαίτερα συναισθηματικά και είναι και θέμα αρκετών αναφορών και ερωτήσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που λαμβάνονται από τους πολίτες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η θερινή ώρα ρυθμίζεται από την Οδηγία 2084 Πρόκειται για την ένατη οδηγία για τη θερινή ώρα, εγκρίθηκε κατόπιν διαδικασία συναπόφασης και μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο μέχρι το τέλος του 2001. Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν ήταν αυτή η οποία εισήγαγε τη θερινή ώρα στην Ευρώπη, ήταν απλώς ένα μέτρο εναρμόνισης. Η πτυχή της εναρμόνισης αντανακλάται σαφώς στην επιλογή της νομικής βάσης, πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 114 της Ενθικής Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει την έγκριση μέτρων για την προσέγγιση της νομοθεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην ουσία οι περισσότερες χώρες ε, έχουν ε, δική τους ιστορία θερινής ώρας. Η Γερμανία και κάποιες άλλες είχαν ήδη εισαγάγει θερινή ώρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά οι περισσότερες χώρες αναβίωσαν τη θερινή ώρα κατά τη δεκαετία του 70 και του 80. Κυρίως έγινε για τρεις λόγους. Ένας ήταν η εξοκοινόμηση ενέργεια ε, στη δεκαετία του 70 να υπενθυμίσω ότι είχαμε και την πετρελαϊκή κρίση. Επίσης θέλαμε να υπάρχει περισσότερο φως ε, τα απογεύματα ώστε να υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες να μπορεί να γίνουν μετά τη δουλειά ή μετά το σχολείο. Επίσης ε, μπορούμε να έχουμε ένα ε, πρόγραμμα ταυτόχρονης ώρας με γειτονικέ χώρες που επίσης βοηθούσε τα κράτη-μέλη. Και φυσικά αυτό συμπεριλήφθηκε στην Εθνική Νομοθεσία. Στην αρχή τα κρατη μελη τηρούσαν τη θερινή ώρα με δικό τους πρόγραμμα και αυτό θεωρήθηκε πρόβλημα για την εσωτερική αγορά, κυρίως για τις διασυνοριακές μεταφορές, τις επικοινωνίες και το εμπόριο. Η πρώτη απόπειρα εναρμόνισας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 1975, αλλά χρειάστηκαν 25 χρόνια και 9 οδηγίες προκειμένου να έχουμε πλήρη ευρωπαϊκή εναρμόνιση ε, για τη θερινή ώρα. Ε, να σας πω δύο λόγια και για το διεθνές πλαίσιο. Σήμερα η θερινή ώρα τηρείται σε πάνω από 60 χώρες παγκοσμίω ε, και κυρίως ε, στο βιομηχανοποιημένο κόσμο, στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη και σε κάποιο βαθμό και στη Μέση Ανατολή. Στην Ευρώπη μόνο τέσσερις χώρες δεν εφαρμόζουν θερινή ώρα. Η Ισλανδία, η Λευκορωσία, η Ρωσία και η Τουρκία. Όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλάζουν τα ρολόγια τους και μάλιστα συγχρονισμένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι χώρες που το κάνουν στην Ευρώπη επίσης τηρούν τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες και ερευνητικά έγγραφα που εξετάζουν τις διάφορες πτυχές της θερινής ώρας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις πιθανές συνέπειες για διάφορους οικονομικούς τομείς και την υγεία ε, σε αρκετές εξωτερικές μελέτες. Το 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αξιολόγηση επιπτώσεων για να υπάρχει ενημερωμένη νομοθετική πρόταση για την παρούσα οδηγία του 2000 μετά το 2007 ε, υπήρξε μια έκθεση παρακολούθησης για να ελέγξουμε κατά πόσον η υπόθεση του 2000 εξακολουθεί να ισχύει. Η έκθεση αυτή ζητήθηκε από την ίδια την διάταξη της οδηγίας. Το Γραφείο Τεχνολογίας στο γερμανικό Bundestag, το οποίο συμβουλεύει το γερμανικό κοινοβούλιο, το Bundestag, για θέματα τεχνικών και επιστημονικών αλλαγών, χρησιμοποίησε αυτή τη μελέτη ως σημείο αφετηρίας για μια μεγάλη έρευνα. Τα πορίσματα δημοσιεύτηκαν ε, την άνοιξη του 2016. Αυτή είναι η πληρέστερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ για το θέμα αυτό. Το έργο εξέτασε τα στοιχεία που υπάρχουν, είτε επιστημονικά είτε μη, τα οποία έχουν δημοσιευθεί από το 2007 και τούδε, και έκανε σύγκριση με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007. Αυτό το οποίο ε, προσδίδει μεγάλη αξία σε αυτή την έκθεση είναι ότι αναλύει ε, διεξοδικά και τη μεθοδολογία που αφορά οποιοδήποτε ερευνητικό ε, έγγραφο. Και πολύ συχνά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και οι εξωτερικοί παράγοντε μπορούν να εξηγήσουν γιατί υπάρχουν διάφορε μελέτε οι οποίε καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Η μελέτη του EPRS έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης του Bundestag και Τη συμπληρήσαμε με σχετικά πορίσματα, ε, τα οποία έχουν δημοσιευθεί ε, εντωμεταξύ σε ερευνητικά έγγραφα. Εξετάζει την κατάσταση στην εσωτερική αγορά φαντάζομαι ε, από εκεί και πέρα και κάθε πτυχή ασφάλειας, υγείας ε, και πολιτιστική πτυχή. Ε, λόγω έλλειψης χρόνου θα επικεντρωθώ στην εσωτερική αγορά και στην ενέργεια και στην υγεία. Όπως σας είπα, κυρίως μας απασχολεί η εσωτερική αγορά, γιατί όπως είπα προηγουμένως, ο βασικός στόχος ήταν η αγαστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η καλή λειτουργία της οδηγίας για τη θερινή αγορά, η ώρα συγγνώμη, στην εσωτερική αγορά μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το κόστος λόγω έλλειψη εναρμόνιση μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το θέμα αυτό σε μια μελέση που έγινε το 2014 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν δεν υπήρχε συγχρονισμός θα υπήρχε υψηλότερο κόστος και χαμηλότερη παραγωγικότητα στην εσωτερική αγορά. Όσο αφορά την ενέργεια, έγιναν έρευνες για το κατά πόσον υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας και είναι μεικτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα από μια χώρα δεν μπορούν πάντα να θεωρηθούν ότι ισχύουν και για άλλη χώρα λόγω γεωγραφικής θέσης ή και συγκεκριμένων συνθήκων ή και νοοτροπίας και πολιτιστικών ε, συνηθιών. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούνται κλιματιστικά ή όχι. Ε, υπάρχουν δύο ενδιάμεσε μελέτες που καταλήγουν ότι όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, κάποιες εξοικονομίες ενέργειας για τα νοικοκυριά, αλλά όχι για τη βιομηχανία. Και η μία μεγάλη τσέχικη μελέτη από το 2016 διαπιστώνεται ότι η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι 0,34% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το φάσμα της υγείας ε, και θέματα που αφορούν τη θερινή ώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν ε, βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στέχοι και πιθανές αρνητικές συνέπειες. Ε, κάποιες μελέτες αναφέρονται στα ωφέλη ε, υπό την έννοια ότι ο κόσμος ε, ε ωφελείται από τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας γιατί κάνει δραστηριότητες στην Ήπεθρο και η άσκηση θεωρείται καλή για την σωστή φυσική κατάσταση και φυσικά το φως του ήλιου είναι απαραίτητο για πρόσληψη βιταμίνης ε, D. Αλλά αυτό το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως επιχείρημα για τη θερινή ώρα είναι το γεγονός ότι διαταράσσονται οι ανθρώπινοι βιορυθμοί, ε, οι κυρκαδιανοί κύκλοι όπως αποκαλούνται. Και αυτό ε, είναι συγκρίσιμο με ένα μικρό jet lag, δηλαδή αυτό που νιώθουμε όταν ταξιδεύουμε μεταξύ διαφορετικών ζωνών. Ε, η διαταραχή και η στέρηση του ύπνου ε, έχουν αποτέλεσμα στη συγκέντρωση και μπορεί να δημιουργήσουν και αϊπνία και ζαλάδα. Ε, πιστεύετε ότι χρειάζονται μερικές μέρες να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα στις αλλαγές, αλλά τα απορίσματα της ανθρώπινης βιολογίας διαπιστώνει ότι διαταράσσεται το βιολογικό ρολόι πολύ λιγότερο από ό,τι πιστεύετε και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσαρμόζονται εύκολα ή δεν προσαρμόζονται καθόλου. Η διαταραχή για το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι κατά πάσα πιθανότητα δέχεται όθηση διότι ε, το φετινό Νόμπελ για την ιατρική ε, δόθηκε σε τρεις ε, Αμερικανούς ερευνητές οι οποίοι ερεύνησαν ακριβώς τους κυρκαδιανούς κύκλους. Και τώρα θα περάσω στην κοινή γνώμη. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο κράτος μέλος το οποίο να έχει ζητήσει αλλαγή ε, του συστήματος, αλλά υπάρχουν αρκετές αναφορές πρωτοβουλίες των πολιτών και πρωτοβουλίες στα εθνικά κοινοβούλια που ζητούν κατάργηση της θερινής ώρας ή της αλλαγής της ώρας. Ε, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι φωνές, ε, υπάρχει ένα κενό γνώσης ε, από πλευράς κοινή γνώμης, διότι η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 90 και του 80 που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τα μισά μέλη και ήταν τελείως διαφορετική η γεωγραφική κατανομή, είναι οι τελευταίες εκδήσεις που έξουμε. Υπάρχουν κάποια ε, που δείχνουν ότι ο κόσμος γενικά είναι πολύ δυσαρεστημένος, κυρίως στη Γερμανία και υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες ε, σε εθνικό επίπεδο, στα κοινοβούλια, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς ξέρουμε ελάχιστα για τη στάση των πολιτών οι οποίοι δεν εκφράζουν την άποψή τους. Είναι ικανοποιημένοι με μεγαλύτερε ε, ε, βραδιές ηλιοφάνειας είναι δυσαρεστημένοι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ε, προτιμούν αλλαγή, προτιμούν να υπάρχει θερινή ώρα κάθε χρόνο ή η συνήθις ώρα κάθε χρόνο. Αυτό δεν είναι σαφές. Κάθε επιλογή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και πριν, ε, συγγνώμη μπορώ να έχω ένα λεπτό ακόμα, ωραία σας ευχαριστώ. Πριν αποφασίσουμε για το ποιο, πρόγραμμα θα, ποιο σύστημα θα ισχύσει, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βασικά ωφέλη και τι συνέπειες θα έχουν η θερινή ή συνήθις ώρα ε, για την ε, Ανατολή και Δύση του ηλίου. Αυτά τα χρονικά περιθώρια σίγουρα μπορούν να ποικίλουν από τη μία χώρα στην άλλη και ανάλογα με την ε, ζώνη στην οποία βρίσκεται η κάθε χώρα, πού είναι τοποθετημένη και το γεωγραφικό πλάτος. Ε, στη μελέτη μας αυτές οι διακυμάνθεις ε, φαίνονται με διαγράμματα. Ε, έχουμε την Αθήνα, τη Βιέννη και τη Στοκχόλμη και υπάρχει και ένα πίνακα στο παράρτημα που περιλαμβάνει στοιχεία για όλες τις χώρες. Και βάσει της παρούσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αποφασίσουν opt-out από την οδηγία, γιατί είναι παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οποιαδήποτε αλλαγή του ε, συστήματος ε, θα απαιτεί αλλαγή της ε, νομοθεσίας, της οδηγίας. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λύσεις. Ή να διατηρήσουμε το status quo, να ανακληθεί η οδηγία ή να τροποποιηθεί. Όσον αφορά την ανάκληση της οδηγίας, επειδή τα κράτη-μέλη έχουν ήδη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, η ανάκληση δεν θα σημαίνει αυτόματη λήξη της θερινής ώρας, θα σταματήσει η εναρμόνιση και η αρμοδιότητα για τη θερινή ώρα, από εκεί και πέρα θα επαφείται στα κράτη-μέλη. Ε, Όσον αφορά την οδηγία για τη θερινή ώρα, τα κράτη-μέλη μπορεί να αποφασίσουν να μην διατηρήσουν ε, την θερινή ώρα ή να μην διατηρήσουν το πρόγραμμα. Έτσι, ροχεύει ο κίνδυνο κατακαιρματισμού, ο οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε στρεβλώσει τη εσωτερική αγορά, ε, προβλήματα για του πολίτε και για τι επιχειρήσει. Τροποποίηση μπορεί να σημαίνει ότι θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να έχουν ένα σύστημα opt-out. Αυτό υπάρχει στι ΗΠΑ, αλλά ελάχιστε πολιτείε το χρησιμοποιούν και κάποιοι προτείνουν να τροποποιηθεί η κείμενη νομοθεσία ώστε η αλλαγή της θερινής ώρας να καταργηθεί πανευρωπαϊκά ε, ε, για όλους. Ε, σε αυτό το σενάριο όμως θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα σημαίνει αυτό για την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου σε κάθε χώρα για να μπορέσουμε να μετριάσουμε οποιασδήποτε ε, παρενέργειες, ε, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει ε, βάσει και της ζώνης στην οποία βρίσκεται. Δεν θα κρίνει βέβαια το EPRS τις μελλοντικέ λύσεις. Η μελέτη έγινε απλώς για να καταλάβουμε με ποια λογική δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται η οδηγία του 2000 και να εξετάσουμε και τις διαθέσιμες επιστημονικές ενδείξεις στους διάφορους τομείς που αφορά η θερινή ώρα. Η μελέτη λοιπόν του EPRS προσπαθεί απλώς να δώσει μια αμερόληπτη συνεισφορά στη συζήτηση. Ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας και συγγνώμη που μακρηγόρησα λίγο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Πολλά καινούργια πράγματα τα οποία δεν τα είχα ήδη καθόλου σκεφτεί. Για παράδειγμα, τι καταστροφή θα ήταν να ε, επιστρέψουμε τις αρμο, την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη. Θα καταλήγαμε σε ένα πλήρες χάος. Κάποιοι θα τεφάρμοζαν την αλλαγή ώρας, κάποιοι όχι. Περνάμε στην ε, αναφρά 2558 ε, για την κατάργηση της αλλαγής ώρας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρον είναι εδώ και θα του δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μ' αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα. Ε, πολλοί όμως εγκαταλείπουν τον αγώνα απέναντι στις, στη γραφειοκρατία των ε, Βρυξελών ε, και η αλλαγή της ώρας αποτελεί λάθος απόφαση σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους. Είναι σύμβολο της κακής γραφειοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί πολίτες ε, θα είχαν ε, περισσότερο σεβασμό απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είχε τη μεγαλοψυχία να πει ότι ναι, δεν ήταν πολύ καλή ιδέα να το αλλάξουμε αυτό. Ε, η αλλαγή Τη ώρα έχει πολλές αρνητικέ συνέπειε. Ε, η μεγαλύτερη ε, ε, ζημιά φαίνεται δύο εβδομάδες μετά κάθε αλλαγή της ώρας, όπου είναι σαφώ αποδυναμωμένοι οι άνθρωποι. Και έτσι βρισκόμαστε σε αντιγωνισμό σε σχέση με χώρες που δεν αλλάζουν ώρα, που δεν έχουν θερινή ώρα και υπάρχουν και οι άμεσες συνέπειες. Τα παιδιά χρειάζονται ύπνο και όταν ε, έχει περισσότερο φως το βράδυ ε, πηγαίνουν πιο αργά για ύπνο. Ε, επίσης, μειώνεται η αποδοτικότητα και η δυνατότητα μάθησης. Όταν έχουμε πολιτικές αποφάσεις, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι, αλλά όσον αφορά την αλλαγή της ώρας ε, οι περισσότεροι δεν είναι ικανοποιημένοι και το πρόβλημα είναι η αλλαγή της ώρας ε, διότι κάποιοι προτιμάνε τη θερινή και κάποιοι προτιμούν ε, την χειμερινή ώρα. Εγώ προτείνω έναν συμβιβασμό να εισαχθεί μια κεντροευρωπαϊκή συμβιβαστική ώρα. Έτσι κανένας δεν θα έχει ακριβώς αυτό που θέλει αλλά κανένας δεν θα είναι τελείως ανικανοποιητός. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο Björklund από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει σουηδικό όνομα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον αναφέροντα. Ε, είμαστε ενήμεροι όλων των αναφορών και είναι αρκετές αυτές που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υπηρεσία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την, ε, αυτόν απολογισμό, την καταγραφή όλων των ε, ερευνητικών αποτελεσμάτων για το ίδιο θέμα. Ε, αναφέρατε και το ιστορικό αυτής της οδηγίας. Ποτέ δεν ήταν στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κομισιόν να ε, εισάγει την καλοκαιρινή ώρα. Ο στόχος ήταν η εναρμόνιση των διαφορετικών καθεστώτων θερινή ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Έτσι κι αλλιώς οι αντίστοιχες αποφάσεις ε, ε, αφορούν τα είναι αρμοδιότητα των κρατών μαλλών. Έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις ζώνες ε, ορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντήσαμε και σε ερώτηση του μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το ίδιο θέμα και έχουμε επιβεβαιώσει ότι το εξετάζουμε το ζήτημα. Εξετάζουμε όλα τα στοιχεία, τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εξετάζουμε τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη και προφανώς ακούμε πολύ προσεκτικά και τη γνώμη των πολιτών μας. Οπότε αυτή η έρευνα της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου είναι ένα πρόσθετο στοιχείο Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα τη λάβουμε υπόψη μας. παράλληλα με τις αναφορές και τις ε, απόψεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε υπέρ μιας ε, συζήτησης που θα γίνει επί τη βάση επιστημονικών στοιχείων. Ευχαριστούμε πολύ και θα εξετάσουμε και θα λάβουμε υπόψη μας και αυτή την έκθεση ε, στις εργασίες μας. Πρόεδρος, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Είπατε ότι το 2017 θα επιστρέψετε ε, με, την με τα αποτέλεσματα της επανεξέτασης. Δεν μένει παρά 1,5 μήνας για το... μέχρι το τέλος του 2017. Πότε μπορούμε να περιμένουμε τα απορίσματά σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω σήμερα πότε θα τελειώσει. Γνωρίζω τη δέσμευσή μας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα ολοκληρωθεί η ε, μελέτη μας. Γνωρίζουμε τι είχαμε πει, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι ε, για το πότε ακριβώς θα τελειώσουμε. Ε, τα είχε, το είχε πει και ο Επιτρόπος Μπούλς τον Οκτώβριο του 2016. Ε, σε αυτό αναφέρομαι. Είχα, είχε πει ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα έχει τελειώσει η εξέταση. Προφανώς όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, οπότε ας πάρουμε την κατάσταση ως έχει, την αφήσουμε ως έχει. Ανοίγω το... Ε, δίνω το λόγο στη συνάδελφη, στην κυρία Άουκεν, καταρχήν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θερινή ώρα. Και θυμάμαι, είμαι αρκετά μεγάλη να θυμάμαι πότε εισήχθηκε για πρώτη φορά. Γεννήθηκαν και τα δύο παιδιά μας περίπου εκείνη την εποχή. Και δυσκολευόμαστε να τα βάλουμε για ύπνο να κοιμηθούν το απόγευμα γιατί ο ήλιος ήταν ακόμα ψηλά. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Στη Δανία τουλάχιστον είναι πολύ καλό. Αν ήμουν Στη Φιλανδία έτσι κι αλλιώς εκεί το καλοκαίρι ο ήλιος δεν δει σχεδόν, αλλά στη Δανία που είναι πιο νότια, που η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα, ε, είναι πολύ ωραίο να έχουμε χειμερινή ώρα, έθερνη ώρα. Ακόμα και η βία στους δρόμους έχει αυξηθεί τώρα πια. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία δεν αλλάζει. Ώρα. Ο, ε, ε, και η Πορτογαλία έχει την ώρα του Greenwich ε, ενώ η, Ισπανία έχει την κεντρική ώρα επειδή ο Φράγκο ήθελε να μιμηθεί το Χίτλερ και οι άνθρωποι πηγαίνουν τα, διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας συνεχώς και έχουν διαφορά ώρας. Και ελπίζω ότι θα διατηρηθεί η θερινή ώρα. Τα προβλήματα δραματοποιούνται νομίζω, μεγαλοποιούνται, μεγενθύνονται. Ε, τώρα με τις αγελάδες, ε, τι διαφορά έχει. Το μόνο που με λυπή είναι ότι καθυστερούμε να επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα. Οπότε ε, δεν χαιρόμαστε τα πιο μεγάλα πρωινά. Θα ήθελα να έχω μία ώρα παραπάνω, λίγο χρόνο παραπάνω το πρωί το χειμώνα. Όμως καθυστερεί η αλλαγή. Ε, δεν, με αυτόν τον ε, τρόπο ε, δεν εποφελούμαστε παρκώς των πρωινών μας το, στην αρχή του χειμώνα. Pork and Bess, ε, θυμάστε το τραγούδι Summer time and the living is easy. Ε, την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψα ότι στο Κοινοβούλιο, όπως και στο Τρασβούργο. Έχουμε τους ε, παλιούς λαμπτήρες πυράκτωσης, ναι, το 150 βάτια παράδειγμα. Οι Φιλανδοί φίλοι μου λένε ότι πια έχουμε LED. Θα έπρεπε να αλλάξουμε τους λαμπτήρες και να τους κάνουμε LED. Όμως εδώ στο Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει τους λαμπτήρες ε, ε, LED. Είμαστε ακόμα στο 19ο αιώνα, Έντισον κλπ. Should Ναι, πολλά λάθη θα πρέπει να διορθωθούν. Πίτερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους ε, αναφέροντες. Ε, πολύ καλή η πρόταση του αναφέροντος ε, Κανεί ε, να μην αποκτήσει αυτό που θέλει τελικά. Αυτό είναι συμβιβασμό. Αν ε, το είχαμε και αυτό στο Βερολίνο θα είχαμε και κυβέρνηση σήμερα. Όσον αφορά τη θερινή και τη χειμερινή ώρα, αυτό που εκνευρίζει περισσότερο τον κόσμο είναι η αλλαγή της ώρας. Όταν μιλώ με τους ε, ψηφοφόρους μου, η αλλαγή της ώρας εκνευρίζει, ενώ το υπόλοιπο δεν τους νοιάζει και υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που λέει αν θα μπορούσαμε να μην έχουμε την αλλαγή της ώρας, να έχουμε απλά θερινή ώρα, αυτό θα ήταν ε, εντάξει. Η μελέτη έδειξε ε, πολύ ωραία ότι σκοπός ήταν η εξοικονόμηση της ενέργειας. Στο μεταξύ όμως υπάρχουν ε, Στο μεταξύ ε, έχουν ε, ε, αναιρεθεί τα επιχειρήματα αυτά, διότι φαίνεται ότι οικονομικά δεν υπάρχει κέρδος. Εάν όμως τώρα θέλουμε να καταργήσουμε την θερινή ώρα, θα υπάρξουν κάποιες άλλες πτυχές και θα ήθελα να επισημάνω πρώτον ότι δεν θα ήθελα κι εγώ να χάσουμε την εναρμόνιση λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην έχουμε μια λύση password. Διότι αυτό θα ήταν καταστροφικό. Ε, ζητώ όμως περισσότερη τόλμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ε, δεν, υπάρχει, δεν είναι μόνο οι αναφέροντες, υπάρχει και ψήφισμα της ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρχε μια ομάδα δράσης που θέλει να αποφύγει την αλλαγή τη ώρα. Εγώ θα ήθελα περισσότερη τόλμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να αλλάξουμε την ώρα ή και όχι. Αλλά πάλι κλείνει το θέμα χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Να υποβάλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λύσουν το πρόβλημα. Να διατηρηθεί φυσικά η εναρμόνιση. Αλλά να εφαρμόσουμε ενιαία ώρα και βέβαια τα κράτη-μέλη θα πρέπει τότε να πάρουν θέση. Ε, στη Γερμανία <laughs> ε, έχουμε και όρο για αυτή τη συμπεριφορά ότι ε, ναι, ναι εντάξει άμα θέλεις αλλά δεν ξέρω και, και λοιπά ε, το 2017 υποτίθεται ότι θα είχαμε ένα αποτέλεσμα από την Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει όχι όμως ας μην βιαζόμαστε. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν, υποβάλλεται επιτέλους μια πρόταση για να πάρουν θέση τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που στο μεταξύ η νομική υπηρεσία έχει ξεκαθαρίσει ποιος μπορεί να κάνει τι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, εάν θέλει, μπορεί να τροποποιήσει την οδηγία. Θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και κατόπιν έχουμε απλά την κανονική νομοθετική διαδικασία. Προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Θα ήθελα να καθησυχάσω και τον ε, αναφέροντα. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει κανεί του νόμου τη φύση, αλλά του ε, νόμου των ανθρώπων ε, μπορεί, μπορεί να του αλλάξει κανεί. Η αλλαγή της ώρας είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, να μην ε, καταλήξει στο δίλημα χειμερινή ή θερινή ώρα, αλλά να πει πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την αλλαγή της ώρας. Και εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ να έχουμε για πάντα τη θερινή ώρα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ για την αναφορά σας. Μας ε, δίνει την αφορμή να συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και ζητώ περισσότερη τόλμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στα κράτη-μέλη ώστε να πάρουν επιτέλους θέση. Και μία τελευταία παρατήρηση. Πολύς χρόνος χρειάστηκε μέχρι να συμφωνήσει η Ευρώπη. Να συμφωνήσουμε πότε να αλλάζουμε την ώρα. Και βέβαια θέλουμε να αποφύγουμε να χαλάσουμε τελείως την κατάσταση. Αλλά μπορεί να, να έχει έρθει η ώρα για την Ευρώπη. Εγώ πάντως θα προτιμούσα θερινή ώρα για πάντα, λέει ο, ο, ο κύριος Γιάρ. Ελπίζω η πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, να συμφωνήσει με την πρόταση αυτή, να έχουμε και ένα ψήφισμα και να ξανασυζητήσουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά από ό,τι φαίνεται οι οικονομικοί λόγοι δεν υπάρχουν πια για την αλλαγή της ώρας. Πολιτικές στοιχές υπάρχουν. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν να ακούσουμε τους πολίτες και να αποφασίσουμε ποια ώρα θα ήταν τελικά η πιο κατάλληλη. Thank you very much, Peter. Ευχαριστώ, Πίτερ. Θα δώσω και πάλι πίσω το λόγο στον κύριο Σάρφερ Νόρτ. Danke. Ähm, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θα ήταν φυσικά πάρα πολύ ωραίο αν γρήγορα είχαμε κατάργηση της αλλαγής της ώρας. Σας ευχαριστώ. I thank you for having traveled all the... Σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Περιμένουμε ανυπόμονα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό διότι το 2017 πλησιάζει στο τέλος του. Εγώ μάλλον αρχές του επόμενου έτους θα περίμενα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιμένουμε ανυπόμονα την πρότασή σας. Ας κάνουμε το εξής λοιπόν, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να περιμένουμε το αποτέλεσμα της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του θέματος αυτού. Νομίζω ότι αυτό ε, συνάδει απόλυτα με αυτά που είπε και ο Πίτερ και σας διαβεβαιώ ότι εδώ στο κοινοβούλιο μας ε, είναι καυτό θέμα. Τόσοι συνάδελφοι έχουν έρθει σε μένα από διάφορες ομάδες πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ προσωπικά ταξιδεύω τόσο πολύ σε όλο τον κόσμο και ζω συχνά αλλαγέ ώρα 7-8 ώρων που η μία ώρα δύο φορές το χρόνο δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι κάτι που απασχολεί περισσότερο άλλους. Ας ε, περιμένουμε λοιπόν ε, την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα τον αναφέροντά μας. Επιστρέψτε στην Γερμανία και να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε κατά νου την αναφορά σας και τις 18 αναφορές για το θέμα αυτό. Υπάρχουν αναφορές όμως και από την άλλη πλευρά. Και ευχαριστώ θερμά και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αποχωρήσω από την αίθουσα τώρα. Θα με αντικαταστήσει ο Παλ Σάκη, αντιπρόεδρός μας. Καταφτάνει, ε? Α, είναι ήδη εδώ. Ωραία. Σύντομο διάλειμμα, θα είναι σύντομα μαζί σας. Και τώρα θα περάσουμε στις τελευταίες δύο αναφορές. Θα ξεκινήσω με την αναφορά 2664 του 2013 του Γκαπριέλ Ζιέο Μπιάνκ. Εξ όσων γνωρίζω δεν είναι εδώ αναφέρον. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Μπαλμαρί ή την κυρία Μπάριος, να μας ε, κάνουν την παρουσίασή τους. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ. Δεν είναι εδώ αναφέρον και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Είναι κάποιος εδώ. Oh, uh, Α, είστε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. από πλευράς υπηρεσία εξωτερική δράσης ε, κάποιες παρατηρήσεις ε, για το γενικότερο πλαίσιο της αναφοράς και μία σύντομη ενημέρωση για το πού βρίσκονται τα πράγματα από τότε που ε, έγινε η αναφορά το 2013 και μετά από την τελευταία συνεισφορά μας το 2015. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική κατάσταση στην σημερινή Γουινέα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες δεν έχει βιώσει κάποια τεράστια αλλαγή ε, και το καθεστώς από το 1990 και πιο πρόσφατα ξεκίνησε ένα πολιτικό άνεγμα υποτίθεται το οποίο όμως δεν έχει οδηγήσει σε κάποια αλλαγή στην εξουσία και η εικόνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ε, ελευθερίες εξακολουθεί να είναι ζωφερή. Όπως ξέρετε υπάρχουν ε, συχνές εκθέσεις από διεθνούς οργανισμούς που αναφέρουν τα σχετικά. Η κατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων, ε, της πολιτικής γνώμης και πολιτικής ελευθερίας αποτελούν σημείο ανησυχία. Κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να είναι στην εξορία ε, και δεν έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές. Κάποια πράγματα τώρα πιο συγκεκριμένα όσον αφορά ε, τους ανθρώπους που αφορά η Επιτροπή. Να πω ότι ο Σεβενούτο, ιστορικό ιστορικό ηγέτης ε, της αντιπολίτευσης, βρίσκεται στην εξορία, έκανε κάποιες διαπραγματεύσει για να επιστρέψει στο Μαλαμπού, αλλά τελικά δεν υπήρξε κάποια συμφωνία που να το επιτρέψει να επιστρέψει από την εξορία και υπήρξαν και κάποια ελιγμοί από το καθεστώς. Ο Γκαμπριέλ Ενσέ, ένας από τους αναφέροντες, ε, κατάφερε να επιστρέψει στην σημερινή ε, Γουινέα, αλλά δεν κατάφερε να ε, δραστηριοποιηθεί στην αντιπολίτευση, γιατί το κόμμα του καταρχάς υπέστη μια σειρά από περιορισμούς και ο ίδιος είναι κατηγορούμενος τους τελευταίους μήνες και βρίσκεται σε κατοίκον κράτηση και δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Τώρα, για να περάσω στις πιο πρόσφατες εξελίξεις που είναι πιο σημαντικές ε, στη πολιτική σφαίρα. Τα γνωρίζετε ότι έγιναν προεδρικές εκλογές το 2016 και η αντιπολίτευση έκανε μποϊκοτάζ στις εκλογές του CPSD, κέρδισε ο πρόεδρος χωρίς να αποτελεί βεβαίως ε, έκπληξη, είναι με 17 χρόνια στην εξουσία. Ε, υπήρχαν ε, κάποια περιστατικά βίας κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Πρόσφατα η ε, χώρα είχε και βουλευτικές εκλογές και δημοτικές εκλογές πέραν των προευρικών. Στις 12 Νοεμβρίου έγιναν αυτές. Οι εκλογές έγιναν γενικά με ειρηνικό τρόπο υπήρχαν κάποιες μικρές ομάδες παρατήρησης από την Αφρικανική Ένωση και κάποια, μια ομάδα πορτογαλόφωνων χωρών, αλλά υπήρχαν ισχυρισμοί για πάρα πολύ σοβαρέ παρατυπίε στις ε, ψήφους της αντιπολίτευσης ε, και ότι το κυβερνών κόμμα ε, θα κερδίσει πάλι με πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως θα είδατε βέβαια και τα αποτελέσματα έδειξαν μια πολύ μεγάλη νίκη του Προεδρικού Κόμματος το οποίο κέρδισε και τις 55 έδρες της Γερουσίας και τις 99 ε, από τις 100 ε, έδρες στην ε, Εθνοσυνέλευση. Αυτά λοιπόν, εν συντομία, εν περιγραφής για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις ε, και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην σημερινή Γουινέα από την τελευταία φορά που ήρθαμε στην Επιτροπή Αναφορών. Να πω επίσης ότι προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ε, συζητά με την κυβέρνηση της σημερινή Γουινέας ε, σε κάθε ευκαιρία προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία τη για την συνολική κατάσταση στην σημερινή Γουινέα και επίσης ενθαρρύνουμε και την ε, κυβέρνηση να λάβει αποφασιστικά βήματα προκειμένου να ε, βελτιώσει την ε, ζωφερή κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική ελευθερία, τον πολιτικό χώρο και γενικότερα την ελευθερία έκφρασης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους αν θα έχουν σχόλια. Όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε προτείνω το εξή για τη συγκεκριμένη αναφορά. Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη, το ζήτημα είναι ε, εξόχως πολιτικό. Η Επιτροπή μας δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση, οπότε προτείνω να στείλουμε μια επιστολή στις Ισπανικές Αρχές, να τις ενημερώσουμε για το πρόβλημα και μια άλλη επιστολή στην κυρία Μογκερίνη, στην οποία θα αναφέρουμε τη συγκεκριμένη αναφορά και το πρόβλημα και μετά από αυτά τα βήματα να κλείσουμε την αναφορά. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε. Βλέπω να συγκατανεύεται. Ωραία. Τελευταία αναφορά που θα εξετάσουμε σήμερα είναι η 0405 του 2017. Ο αναφέρον είναι ο Θέσαρ Δεθφούλη Ρέλιο από την Ισπανία. Έχετε το λόγο κύριε Ρέλιο. Ρέλιο για 5 λεπτά. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε για να σας παρουσιάσω αυτήν την αναφορά που έκανα πριν από αρκετούς μήνες σε ό,τι αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών στη Λιβύη και το εγκλήματα κατά της ε, ανθρωπότητας που λαμβάνουν χώρα σε αυτή ε, την περιοχή. Η, οι μετανάστες υποφέρουν στην ε, Λιβύη και αυτό αποτελεί ε, προσβολή στην, στη ε, συνείδηση ανθρωπότητας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθάει τις λιβυικές, τη να τους επιστρέψουν στην Λιβύη είναι απάνθρωποι. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να κλείνει άλλο τα μάτια. Αυτά δεν είναι τα δικά μου λόγια, αλλά του Σέιτ Ραντ Αλ Χουσέιν, που είναι επικεφαλή τη ε, υπατσαρμοστία του ΟΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι έκανε στι 14 Νοεμβρίου. Πριν από έξι μήνε περίπου ξεκίνησα αυτή την αναφορά ω πολίτη, αλλά και ω δημοσιογράφο. Πραγματικά ήμουν εξοργισμένο εκείνη την εποχή βλέποντα ε, τι ε, εικόνε από τι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα εδώ και αρκετό καιρό τότε θεώρησα, κατάλαβα ότι είναι υποχρέωσή μου να αντιδράσω. Πολλές ε, αποδείξεις ε, ε, έχουν δημοσιευτεί τα, τους τελευταίους μήνες, αλλά και πολλές οργανώσεις, διεθνείς οργανώσεις έχουν καταγγείλει τα γεγονότα. Η Διεθνής Οργάνωση για τους Μετανάστες, τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Αμνηστία, τη Human Rights Watch κλπ. Θα, τα δείτε, θα δείτε επιστολές τους στο, στο φάκελο που έχω υποβάλει. Ε, με υποστηρίζουν πολλές ε, οργανώσεις ε, που δρούν στην Κεντρική Μεσόγειο και τις ευχαριστώ. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Oxfam, η Jugend κλπ. Μερικοί, μερικές από αυτές τις οργανώσεις έχουν στείλει επιστολές. Τα γεγονότα στη Λιβύη απαιτούν να τα προσέξουμε. Διώξεις, υποχρεωτική εργασία, αυθαίρετες ε, συλλήψεις, ε, δολοφονίες, βιασμοί, βασανιστήρια κλπ. Ε, στα κέντρα υποδοχής από δίκτυα λαθρομετανάστευσης. Ακόμα και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας μέσω του πρέσβη στο Νίγηρα αναφέρονται σε αυτές τις πολύ κακές συνθήκες. Περίπου 500.000 ε, μετανάστες ε, έχουν εντοπιστεί στην ε, Λιβύη από τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης. Μετανάστευση. Ναι. Μπορεί πλέον να, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ακόμα περισσότεροι. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που βρίσκονται μέσα σε μια αγορά σκλάβων. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν αποδειχθεί από το CNN πρόσφατα που δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με δημοπράτηση ανθρώπων στη Λιβύη τελευταία. Το 74% των ε, μεταναστών έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια ή έχουν δολοφονηθεί. Ε, σύμφωνα με την έκθεση της Oxfam της 9 Αυγούστου 2017. Δύο μαρτυρίες θα σας διαβάσω. Ο Τσίντι, 18 ετών από την Γκάμπια, μιλάει για τα βασανιστήρια τα οποία ζησε στη Λιβύη. Όταν έφτασα στη Λιβύη το 2016, ε, μια συμμορία με έφερε στην ε, φυλακή Ζουφάρα, ε, όπου περίμενα τρεις μήνες. Τρώγαμε μόνο μια φορά τη μέρα. Και τακτικά ασκούσαν βία πάνω μας και με βασάνιζαν επανειλημμένως με κρέμασαν ως βασανιστήριο ε, από τα χέρια και με έδραναν συνεχώς το κεφάλι. Τζουντ, 25 ετών από την Ιγυρία, που ταπεινώθηκε επανειλημμένο στην ε, τη του. Οι φύλακες ε, ε, μας έδιναν τροφή από μια χαραμάδα στην πόρτα. Πολύ συχνά μας τάπιναν και μας τιμωρούσαν ε, μας άφηναν γυμνούς, μας τραβούσαν από τα αυτιά. Ε, πολύ συχνά μας ανάγκαζαν να ξαπλώσουμε και μας έδερναν. Πολλοί τραυματίστηκαν ε, σοβαρά, ενώ άλλοι χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Πολλοί από αυτούς δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Το 2016 πάνω από 180.000 ε, πήραν το δρόμο για την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου αυτό το κοινοβούλιο σας όπως και άλλα ε, αν ε, ε, ε ενέκριναν την κατάρτιση της ακτοφυλακής της Λιβύης και της κυβέρνησης της Λιβύης προκειμένου να σταματήσουν αυτοί το, τις ροές. Τρεις κυβερνήσεις έχει η χώρα και προφανώς καμία από αυτέ ε, δεν ελέγχει το, όλη την επικράτεια. Θέλω να ρωτήσω, είναι δυνατόν να δίνουμε υπεργολαβία την ε, προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αντιληπτό ότι τα χρήματα που δίνουμε στην κυβέρνηση της Λιβύης ε, προορίζεται για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Μπορεί ε, να το κοινοβούλιο σας ε, να είναι συνένοχο σε μια τέτοιου χρηματοδότηση. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν να παραβαίνουν τις διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση αυτή για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Η ακτοφυλακή της Λιβύης σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξασφαλίζεται η επιστροφή στην σε ασφαλή σημεία των προσφύγων οι οποίοι ε, συλλαμβάνονται από την Λιβιακή ακτοφυλακή. Πολλές μαρτυρίες ε, αναφέρουν την εξαιρετικά κακή κατάσταση των επιστρεφόμενων προσφύγων στα στρατόπεδα στη Λιβύη. Επίσης να σας πω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που κάνουν διάσωση στη θάλασσα και τις οποίες διώκει η Ιταλική κυβέρνηση έχουν κάνει ε, ε, έχουν διαπιστώσει ε, επιθέσεις τον Λιβικό της Λιβικής Ακτοφυλακής που οδήγησαν και σε θανάτους. Όσοι, ε, όσοι θα διασωθούν φέτος και θα μεταφερθούν στην Ιταλία είναι λιγότερα από πέρσι. Ε, οπότε ο στόχος έχει επιτευχθεί, αλλά με τι κόστος. Είναι λογικό, είναι νόμιμο να μπλοκάρουμε αυτή την δίωδο διαφυγής των μεταναστών. Προφανώς κανείς δεν θέλει ε, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή του ε, στη θάλασσα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε και αυτοί οι μετανάστες να βρίσκονται σε κίνδυνο στην, ε, στη Λιβύη. δεν υπάρχει κανείς εκεί να διαπιστώσει το θάνατό τους στη θάλασσα, αλλά ούτε και στην, στα τόπεδα στη Λιβύη. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση που χρειάζεται πολιτικέ απαντήσει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη τη ε, Λισαβόνα περιλαμβάνει τι θεμελιώδει αρχέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία κλπ. Ε, δεν ε, είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε στην ειρήνη και στην, στο σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Καλό το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει κατάλληλε έρευνε που να διευκρινίσουν το τι σημαίνει στη Λιβύη σχετικά με τι συστηματικέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον μεταναστών. Θα πρέπει να θέσουμε ε, σε, να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στις ε, συμφωνίες που έχουν ε, υπογραφεί με την Λιβύη. Θα πρέπει να δούμε διεθνείς συμφωνίες έτσι ώστε αυτοί οι μετανάστες να μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους με έναν τρόπο ασφαλή και να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα λαθρεμπόρων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξαναγίνει σημείο αναφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρέγιο. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαν Κρίστοφερ Φίλωρη για να ε, παρουσιάσει ε, την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να ξεκινήσω από μία ενημέρωση για να ε, διευκρινίσω κάποιες παρεξηγήσεις, κάποιες παρανοήσεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, με τους μετανάστες ε, στη Λιβύη όντως ε, είναι επονίδιστο. Τα κέντρα κράτησης στη Λιβύη είναι επονίδιστα. Η ταχύριση των ανθρώπων, το εμπόριο ανθρώπων και η δουλεία την οποία δυστυχώς διαπιστώνουμε και καταγγέλλεται και από πολλά μέσα πρόσφατα είναι μια επίθεση στην ε, ανθρώπινη εξωπρέπεια και στη συνείδησή μας. Επ' αυτόν συμφωνούμε όλοι και συνειδητοποιούμε απολύτως ε, ε, για το επίγον, το επίγον της κατάστασης και γι' αυτό και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Αλλά αυτό το οποίο επίσης είναι υπονοείδιστο είναι και ο αριθμός των μεταναστών που πεθαίνουν στη θάλασσα. 3.771 το 2015, 5.000 το 2016, πάνω από 2.000 ήδη το 2017. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να ξεχνάμε από πού ξεκίνησε η κινητοποίησή μας. Όταν υπήρχαν κάποια σκάφη τα οποία βούλιαζαν στις ακτές της Σικελίας το 2015 και είχαμε πάνω από 800 ναυαγούς και ελπίζω να μην ε, ξεχνάμε ε, και την αγανάκτηση ε, που νιώσαμε εκείνη την ημέρα και που ήταν και αυτή η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τις προσπάθειές μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πολύ σύντομα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν αυτό, γίνονται αυτά τα ναυάγια. Πολλές φορές οι μετανάστες υποχρεώνονται να επιβιβαστούν σε φουσκωτά σκάφη, τα οποία ξέρουμε ότι δεν είναι ε, κατάλληλα για να επιβιώσει κάποιος ε, ε, αυτό το πέρασμα. Είναι εγκληματική η πράξη και επειδή ακριβώς είναι εγκληματική και είναι όνειδος, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και κάτι γι' αυτό και ε, δεν θα πρέπει να συζητούμε καν ε, τους ε, νεκρούς στην έρημο στη Λιβύη, διότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις, αλλά μπορούμε να φανταστούμε και σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχουν πάρα πολλά θύματα. Και φυσικά ε, η κατάσταση ε, σύραξης που υπάρχει στη Λιβύη είναι αυτή η οποία ευνοεί αυτή την τραγωδία που ζουν οι μετανάστες ε, στη χώρα. Και ενώπιον όλων αυτών τι μπορεί να κάνει κανείς. Έχουμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Είπαμε ότι η Λιβύη είναι ε, όντως ένα νεκροταφείο, αλλά δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα, διότι ε, δεν έχουμε πρόσβαση ε, στην απαραίτητη πολιτική μόχλευση για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Και αναρωτιέμαι ποια θα ήταν η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, για παράδειγμα, ε, εάν δεν κάνουμε τίποτα. Η άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι η δεύτερη επιλογή φυσικά, ε, την οποία ε, κάναμε ε, και την επιλογή να ακολουθήσουμε. Και υπάρχει μια στρατηγική για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία. Να σώσουμε τις ζωές αυτών των ανθρώπων, να προστατεύσουμε τους μετανάστες και να σταθεροποιήσουμε τη Λιβύη. Και όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας αυτή τη στιγμή το ε, καταπίστευμα επίγουσας βοήθειας για την Αφρική, το οποίο γεννήθηκε στη Σύνοδο της Βαλέτας ε, το 2015, ε, υλοποιεί στη Λιβύη κάποια προγράμματα που αυτή τη στιγμή ε, αριθμούν εκατομμύρια ευρώ, 162 πιο συγκεκριμένα, 120 εκατομμύρια από αυτά, περίπου τα 3 τέταρτα, προβλέπονται αποκλειστικά για την προστασία των μεταναστών και τη σταθεροποίηση των ε, κοινοτήτων υποδοχής. Τι εννοούμε με τον όρο προστασία. Υπάρχουν ε, ε, ο OIM και η ύπατη ε, αρμοστή για τους πρόσφυγες ε, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μετανάστες στο σημείο επιβίβασής τους, αποβίβασής τους μάλλον από τα σκάφη. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάποιος θα αναλάβει αυτούς τους ανθρώπους. Ο ΟΑΙΑΜ και η αρμοστία βρίσκουν ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι από αυτούς ο ΑΙΕΜ εξασφαλίζει σε αυτούς τους πιο ευάλωτες ε, μετανάστες τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους με ε, ένα οικονομικό πακέτο το οποίο τους επιτρέπει να επανενταχθούν στην κοινωνία. Ο ΑΙΕΜ και ο, η Πατερμοστία για, την, για τους πρόσφυγες δραστηριοποιούνται και στα κέντρα κράτησης και ο στόχος δεν είναι να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στα κέντρα κράτησης αλλά να αποχωρήσουν από τα κέντρα κράτησης και όλες οι προσπάθειες που κάνουν αυτές οι οργανώσεις γίνονται ακριβώς για αυτό το λόγο. Για άλλη μια φορά φυσικά και ε, μέσω των προγραμμάτων εθελοντικής επιστροφής ε, και ένταξης. Και όλα αυτά συνοδεύονται και από μια ε, στρατηγική ε, αμήλικτων πιέσεων προς ε, τις αρχές της Λιβύης, τουλάχιστον αυτών που ελέγχουν τα κέντρα κράτησης ε, στα οποία έχουμε πρόσβαση και πιέσεις λοιπόν ώστε να περάσουμε από ένα μοντέλο κλειστών κέντρων κράτησης σε κέντρα ανοιχτής υποδοχής, σε μάλλον ανοιχτά κέντρα υποδοχής. Ε, από ό,τι άκουσα, ε, θα υπάρξει σύντομα μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μεταβεί στη Λιβύη. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους βουλευτές που θα μεταβούν επί τόπου να διαβιβάσουν αυτό το μήνυμα στις λιβικές αρχές. Ακριβώς για να επιτρέψουμε να έχουμε ανοιχτά κέντρα υποδοχής. Έγινε πρόσφατα ένα πολύ μικρό βηματάκι, ε, διότι οι δύο οργανισμοί ανακοίνωσαν ότι ανοίγει ε, ένα σύνολο ε, ασφαλών χώρων, safe spaces, που επιτρέπουν να ε, τοποθετηθούν οι πιο ευάλωτοι μετανάστες σε οικογένειες υποδοχής, σε κάποιες κατοικίες ή σε χώρους υποδοχής. Είναι ένα μικρό βήμα, α, είναι ακόμα στα σπάργανα, αλλά είναι αυτό το μοντέλο που θα θέλαμε να αναπτύξουμε και να έχουμε στη Λιβύη. Η σταθεροποίηση των ε, κοινοτήτων υποδοχή είναι το επόμενο βήμα. Θέλουμε εκεί να βεβαιωθούμε ότι οι κοινότητε υποδοχέ ε, στους Δήμους θα μπορούν να υποδεχθούν τους μετανάστες ε, με αξιοπρεπείς συνθήκες και να μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα τους παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες και σε Λίβιους αλλά και σε μετανάστες. Και εδώ φυσικά ε, έχουμε ε, κάποιες πιο συνήθεις μορφές υποδοχές, να τους παρέχετε για παράδειγμα ε, νερό, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση ή και υγειονομικό υλικό. Και επίσης είμαστε καθοδόν για να υπογράψουμε με την Ιταλία ένα πρόγραμμα διαχείρισης των συνόρων, το οποίο περιλαμβάνει και διάφορες συνιστώσεις και μία εκ των συνιστωσών είναι ακριβώς ε, να ε, παρέχουμε στην ε, Λιβική Ακτοφυλακή μία πιο επαγγελματική επιμόρφωση από αυτή που έχει αυτή τη στιγμή, διότι αυτή τη στιγμή η Ακτοφυλακή της Λιβύης δεν είναι μια δύναμη που μπορεί να κάνει επαγγελματική διάσωση στη θάλασσα των μεταναστών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να δράσουμε. Να φροντίσουμε, για παράδειγμα, σε περίπτωση που γίνεται διάσωση στη θάλασσα, να την χάνουν αξιοπρεπούς ε, συμπεριφοράς ε, και επαγγελματική συμπεριφοράς οι μετανάστες. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε και τη διακίνηση. Ε, να καταπολεμήσουμε τη λαθρεμπορία και την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων που είναι τμήμα του προβλήματος και από αυτού συμφωνούμε. Και τέλος κάτι ε, τελευταίο. Εμείς δεν χρηματοδοτούμε τη Λιβική κυβέρνηση, δεν ε, χρηματοδοτούμε τις παραστρατιωτικές ομάδες, δεν χρηματοδοτούμε τα κέντρα κράτησης στη Λιβύη. Τα χρήματά μας πηγαίνουν στους εταίρους που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση, για να μπορέσουν να βοηθήσουν απευθείας τους μετανάστες που κρατούνται στα κέντρα κράτησης και να εξασφαλίσουμε και στην τοπική κοινότητα ότι θα υπάρχουν συνθήκες ζωής αξιοπρεπής που θα επιτρέπουν να προστατεύονται και οι μετανάστες. Συνεπώς, με δύο λόγια κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι και αγαπητέ κύριε ε, που υποβάλλεται την αναφορά, αποφασίσαμε να δράσουμε, διότι η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ τον, την Κομισιόν. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Κύριε Αλμπιόλ. Καταρχήν πραγματικά με λυπή που δεν έχουμε μεγάλη προσέλευση ευρωβουλευτών για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Ε, ο αναφέρον μας περιέγραψε μια κατάσταση τραγική Κρίμα που δεν έχουμε περισσότερους ευρωβουλευτές εδώ. Είμαστε επικριτικοί σε σχέση με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από απομακρύνσεις, ε, υπεργολαβή εξωτερική ανάθεση προστασίας των συνόρων, εγκλισμός σε στρατόπεδα κλπ. Ε, και αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα τη κατάσταση που δημιουργεί η εξωτερική ανάθεση τη προστασία των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει μια τρίτη χώρα έτσι ώστε να αναλάβει αυτή η τρίτη χώρα, ε, σαν ανεδεσμοφύλακα, ε, να αναλάβει του ε, μετανάστε. Οπότε περνάμε την ευθύνη σε κάποιον άλλον πληρώνοντά τον. Συμφωνίε με τρίτε χώρε που πολύ συχνά δεν δίνουν εχέγγυα προστασία των δικαιωμάτων. Υπάρχουν συμφωνίες με το Μαρόκο, με την Τουρκία, αλλά ιδιαίτερα αιματηρή είναι αυτή με τη Λιβύα. 160 εκατομμύρια ευρώ ε, σε ένα ειδικό ε, ταμείο για μια χώρα που δεν, χαρακτη... δεν έχει επίσημη κυβέρνηση, είναι ένα κατεστραμμένο κράτος, ερυπωμένο κράτος. Κάποια Κάποιες ε, παραστρατιωτικές ε, ομάδες έχουν ονομαστεί ακτοφυλακή, δεν ξέρουμε, υπάρχουν 7 διαφορετικές ομάδες, δεν ξέρουμε ποια από αυτές είναι οι η ακτοφυλακή και οι 7 ονομάζουν τον εαυτό τους ακτοφυλακή. Ποια από αυτές οι 7 χρηματοδοτείται από εμάς, τι γίνεται δεν ξέρει κανένας. Και βέβαια τα, τους καταβλισμούς ε, κράτησης, ε, πολλοί τους έχουν ονομάσει στρατόπεδα συγκέντρωσης, γίνονται διαδελοφονίες βιασμοί, ε, βασανιστήρια, επικρατούν συνθήκες δουλείας, όλα αυτά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά χρηματοδοτούμε. Αυτά επιτρέπουμε να λαμβάνουν χώρα. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μας ε, θέτει το δίλημα. Ή δούλη στην Λιβύη ή νεκρή στη θάλασσα. Επιλέξτε. Αυτό μας θέτει ως δίλημα η Κομισιόν. Όχι. Δεν είναι αυτή, αυτό το δίλημα. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Μπορεί να δημιουργηθεί μια νόμιμη δίωδος εισόδου προς την Ευρώπη, ε, ασφαλής δίωδος. Μπορούν να δοθούν θεωρήσεις στις πρεσβείες μας έτσι ώστε να φτιάξουν στην Ευρώπη. Το, το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν θέλει να έρθουν στην Ευρώπη. Δεν θέλουν να τους αφήσουν να πατήσουν το πόδι τους στο ευρωπαϊκό έδαφος. Οπότε βέβαια τι μένει, ή θα πεθάνουν στην ε, θάλασσα ή θα ε, εργάζονται 10 χρόνια σαν σκλάβοι και πάλι σε εργοστάσια υφαντουργία στην ε, Τουρκία ή θα μείνουν στους καταβλισμούς εκεί να τους βασανίζουν να τους σκοτώνουν. Λένε, δεν υπάρχει αναλυτική λύση. Και βέβαια υπάρχει αναλυτική λύση. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να φτάσουν με νόμιμο και ασφαλή τρόπο στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών. Δεν είναι η πρώτη αναφορά που μας φτάνει για θέματα μετανάστευσης. Ε, ε, έχουμε αντίστοιχες αναφορές για την Τουρκία και άλλες χώρες. Γιατί, γιατί οι πολίτες μας ανησυχούν. Ήδη ανησυχούν για, τις, ε, τη δράση των κυβερνήσεών μας. Έχουμε πολλού, πολλές οργανώσεις που διοργανώνουν ε, εκδηλώσεις και διαδηλώσεις υπέρ της έλευσης των προσφύγων. Το ακριβώς αντίθετο κάνουν οι κυβερνήσεις μας. Οπότε προτείνω να ενημερώσουμε την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας στείλει όλες οι εκθέσεις που έχει για την εξωτερική ανάθεση των εξωτερικών συνόρων, τι συμφωνίες υφίστανται με τη Λιβύη, τι έχει έγκαια προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι εγγυήσεις ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ λοιπόν η Κομισιόν να μας ενημερώσει, να μας τα στείλει αυτά και να σταλούν επίσης και στον αναφέροντα. Και τέλος, στους συντονιστές θα θέλαμε να εξετάσουμε την περίπτωση, τη δυνατότητα να υποβληθεί μια ε, ε, προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν στην Ολομέλεια. Αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε μεταξύ των συντονιστών. Κάποια όμως αντίδραση, κάποια απάντηση πρέπει να δώσουμε. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ε, μαγνητοσκοπείται η σημερινή συνεδρίαση, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να παρακολουθήσουν ευρωβουλευτές ε, και άλλοι τις συζητήσεις μας. Έχω εδώ γραπτή θέση του ΕΛΚ που στηρίζει την αναφορά σας και προτείνει να παραμείνει ανοιχτή, διότι είναι αναφορά για ένα πολύ σημαντικό θέμα ως πρόεδρος. Ε, εκτιμώ τις ε, δραστηριότητες που περιέγραψε ο κύριος Φιλωρή και επαναλαμβάνω ότι ανέφερε ακριβώς τι χρηματοδοτούμε και τι όχι με ευρωπαϊκούς πόρους. Εγώ βρίσκομαι εδώ σήμερα όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής αλλά και ως εκπρόσωπος του ΕΛΚ και πιστεύω ότι τα προβλήματα ότι δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της Αφρικής και της Ασίας φέροντας όλους τους ανθρώπους εδώ. Είμαστε μια μικρή ήπειρος με περιορισμένους πόρους. Ε, συμφωνώ όμως με τις απόψεις ε, που εκφράστηκαν εδώ ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, θα πρέπει να συμμετέχουμε στην προσπάθεια. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την προσπάθειά του και την αναφορά του. Νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τις προτάσεις ε, των συναδέρφων μου εδώ. Θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε να έχουμε συζητήσεις με τις ε, λιβικές αρχές. Ε, θα, ε, θα στείλουμε ενημερωτικά την αναφορά σας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπως προτάθηκε. Επίσης, θα ζητήσουμε τη θέση της Επιτροπής ΑΦΕΤ, διότι είναι θέμα δικής τους αρμοδιότητας. Και προτείνω, καταρχάς φυσικά, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. και να δούμε ε, σε τι θα καταλήξουν οι συνάδελφοί μας στη Λιβύη. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν θα έχουμε συλλέξει αρκετές πρόσθετες πληροφορίες, θα επανέλθουμε στην αναφορά αυτή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση σε συνεργασία με άλλες επιτροπές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επανέλθουμε στο θέμα. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Συμφωνείτε με την προτινόμενη διαδικασία? Ωραία. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα Συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.